So, uh, αγαπητοί συνάδελφοι. Καλώς ήρθατε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Αρχίζουμε με την ημερήσια διάταξη. Έγκριση της ημερήσιας διάταξη, Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση, θα εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη. Θα ήθελα να καλωσορίσω ένα νέο συνάδελφο στην ομάδα, μα, ομάδα μας που αντικαθιστά τον κύριο Ντάνκαν, ο κύριος Ρούπερτ Μάθιους. Ίσως τον δείτε αύριο, δεν τον βλέπω σήμερα. Προς ενημέρωσή σας αυτό. Μετά, να σας υπενθυμίσω πως έχουμε κάποιες κοινέ συνεδριάσεις με άλλες επιτροπές. Την Τετάρτη, μεθαύριο το πρωί, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για τον, ε, το Κέντρο Συντονισμού Άμεσης Ανάγκης μαζί με την Επιτροπή Ανάπτυξης. Μετά έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων για το track and trace των προϊόντων καπνού με την Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού και με την ίδια επιτροπή μια παρουσίαση του, της ειδικής έκθεσης του ελεκτικού συνεδρίου για τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες απελεγγύε απόψεων, γι' αυτό λοιπόν να σας καλώ να παρευρεθείτε όλοι. Αν και ορισμένοι είστε ήδη εδώ. Τρίτον, έχω καλά νέα για τον Αύγουστο. Στις 30 Αυγούστου, το απόγευμα, Η συνεδρίαση που ε, είχε προγραμματιστεί ακυρώθηκε. Γι' αυτό θα αρχίσουμε στις 31 Αυγούστου, 5η, το πρωί. Και θα ψηφίσουμε μια γνωμοδότηση ε, της Επιτροπής για την Επιτροπή Προϋπολογισμού με αρκετές τροπολογίες. Μετά υπάρχει μια έκθεση της επίσκεψης της Επιτροπής ε, μας ε, στη, στο Λονδίνο, στον EMA, ε, τον Απριλίο, στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων. Μετά έχουμε αποσπασμένους εθνικούς εμπειρογνώμονες που θα φύγουν στις 31 Ιουλίου για να επιστρέψουν στο Υπουργείο τους και εκ μέρους της Επιτροπής Περιβάλλοντος θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Έμπερ για τη δουλειά που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια στην Επιτροπή μας. Και να του ευχηθώ καλή συνέχεια. Είναι εδώ. Εδώ είστε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά, η σημερινή συνεδρίαση θα μεταδοθεί σε 20 γλώσσες και το ηλεκτρονικό αρχείο θα είναι διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής e-meeting. Επίσης, η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο, ζωντανά. Μετά, να εγκρίνουμε τα πρακτικά των συνεδριάσεων της 8ης Ιουνίου και της 12ης Ιουνίου. Εφόσον δεν υπάρχουν ενστάσεις μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, εγκρίνονται. Μετά, περνάμε στο πρώτο θέμα για σήμερα, Γενικό Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό Έτος 2018 θα εξετάσουμε ένα σχέδιο γνωμοδότησης του οποίου ήμουν επικεφαλής ως ε, πρόεδρος μαζί με τους συντονιστές. Θα ήθελα λοιπόν να πω δύο λόγια για το θέμα αυτό. Στις 30 Μαΐου λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε το σχέδιο προπολογισμού το 2018 και εστίασε στις θέσεις απασχόλησης, επενδύσεις, μετανάστευση και την ασφάλεια. Σε γενικές γραμμές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναρμόνισε την πρόταση για το 2018 στα ποσά που προβλέπονται από το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 όπως τροποποιήθηκαν από την ενδιάμεση αναθεώρηση που εγκρίθηκε φέτο. Ο Επίτροπος Ότινγκερ τόνισε ότι το σχέδιο προπολογισμού για το επόμενο έτος ίσως είναι το τελευταίο για τα 28 κράτη-μέλη. Και στο σχέδιο γνωμοδότησης προσπάθησα να τονίσω ότι πρέπει να καταβληθεί κάθε προσπάθεια για να φτάσουμε το στόχο του 20% για κονδύλια που σχετίζονται με το κλίμα καθώς 19,5% των κονδυλίων το επόμενο έτος ε, αφορούν το κλίμα. Και ο προϋπολογισμός έτσι όπως είναι θα δώσει τη δυνατότητα μόνο για 18,5% υπό το φυστάμενο δημοσιονομικό πλαίσιο. Έτσι ώστε να καταναμηθούν λοιπόν οι πόροι και να δοθού, δοθεί έμφαση στην ευγενικότητα και στην προστασία του περιβάλλοντος, να πω ότι Λυπάμαι πολύ για την μείωση του προσωπικού οργανισμών ε, που είναι αρμοδιότητα της Επιτροπής μας ή ε, ε, μείον τρεις θέσεις, Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμα... Χημικών μείον δύο, η CDC μείον δύο θέσεις, ΕΦΣΑ μείον τέσσερις και Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων μείον πέντε θέσεις. Αυτή η μείωση θα επηρεάσει αρνητικά τα καθήκοντα των οργανισμών αυτών, τα οποία αυξάνονται Συνεχώ. και οι οργανισμοί αυτοί θα έπρεπε να διαθέτουν αρκετού πόρου και ανθρώπινο δυναμικό για να εκτελέσουν τι αρμοδιότητές του. Θα υποβάλω λοιπόν σχετικέ τροπολογίε. Τέλο, θα ήθελα να σα υπενθυμίσω ότι τα πιλωτικά προγράμματα και οι προπαρασκευαστικέ δράσει πρέπει να λάβουν επίση επαρκή χρηματοδότηση καθ' όλον τον κύκλο ζωή του, έτσι ώστε να αξιοποιήσουν όλο του το δυναμικό. Ορισμένα πιλωτικά προγράμματα και προπαρασκευαστικέ δράσει, να σα υπενθυμίσω, πως ε, εάν πως ε, εστάλησαν στην Επιτροπή για μία ε, πρώτερη αξιολόγηση. Εάν αυτά συμπεριληφθούν στον προϋπολογισμό και εγκριθούν, πρέπει επίσης να, το, να υποβληθούν ως δημοσιονομικές τροπολογίες μέχρι, τις, μέχρι το τέλος του Ιουλίου. Μετά, το σχέδιο για τον προϋπολογισμό θα είναι διαθέσιμο περί τα τέλη Ιουλίου, από τις 20 μέχρι τις 24 εκτιμώ. Και αυτή είναι και η προθεσμία υποβολής τροπολογιών. Και ε, δεδομένων των θερινών διακοπών, οι τροπολογίες που αφορούν την Επιτροπή Περιβάλλοντος πρέπει να ε, υποβληθούν γιατί είναι θέμα αρχής θέλουν να γίνουν ε, περικοπές και πρέπει λοιπόν να δράσουμε. Αυτά λοιπόν τα λίγα για το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξα. Τώρα θα ήθελα να δώσω σε εσάς το λόγο, αν το επιθυμείτε, και να μου πείτε τις σκέψεις σας και τις απόψεις σας. Θα αρχίσουμε με την ε, κυρία Κάντεμπαχ, η οποία είναι η σκιώδη συγκήτρια από τους Σοσιαλδημοκράτες. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το καλό σχέδιο γνωμοδότησης ενσωματώνει τις ανησυχίες μας. Χαίρομαι που είπατε ότι οι οργανισμοί κάνουν όλο και περισσότερα πράγματα, ε, κάνουν καλή δουλειά και αποδοκιμάζεται τη μείωση προσωπικού. Επίσης, η του προσωπικού τα πρόσφατα χρόνια συμπεριλαμβάνουν και προσωπικό που δουλεύει ε, ε, σε οργανισμούς οι οποίοι χρηματοδοτούνται από τέλη των ετούντων. Δεν συμφωνούμε με αυτό. Επίσης, ε, για το Brexit δεν συμφωνώ. Πιστεύω ότι στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων θα υπάρχει επίπτωση από τον Brexit και ο Οργανισμός Φαρμάκων θα, ε, το 2018 θα έχει επιπλέον φόρτο εργασία λόγω τη απόφασης του Μένου Βασιλείου να αποσυρθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ήθελα να το διευκρινίσω. Α, δεν θέλουμε να υποσκάψουμε το, τις γενικές διαπραγματεύσεις σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των 27 αλλά για να καλύψουμε τις άμεσες ανάγκες του οργανισμού φαρμάκων που χρειάζεται και προσωπικό και χρήματα για να αντισταθμίσει τις απώλειες που θα έχει λόγω του ότι θα αναγκαστεί να μετεγκατασταθεί. Ε, επίσης, Επίση, θα ήθελα παρενθετικά να σα πω ότι καλωσορίζουμε τον ΕΜΑ στην Βιέννη, αλλά αυτό δεν είναι θέμα τη έκθεση βέβαια. Ε, η κυρία Γκάλιν δεν είναι εδώ από το ECR. Από... Η κυρία Αντερμάρκη από τους φιλελεύθερους είναι εδώ. Όχι. Ο κύριος Φλάνναγκαν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ. Πας. Τι έχεις να μας πεις. Όλοι έχουμε διάθεση για διακοπές, έτσι, προφανώς. Ε, ευχαριστώ για την έκθεση, γιατί τα στοιχεία που αναφέρεις ε, τονίζουν ε, τη χρηματοδότηση 20% και την μείωση που, μειώνουμε, που προβλέπουμε για το LIFE. Ε, αναφέρεις και τους οργανισμούς, όλα αυτά που λες για αυτά τα θέματα τα υποστηρίζουμε. Ετοιμάζουμε κάνα δύο τροπολογίες ε, προς την κατεύθυνση αυτών που είπες. Ίσως θα εστιάσουμε περισσότερο στο ότι μπορεί να, ε, με την ε, με το να μην φτάσουμε στο 20% της ε, κλιματικής χρηματοδότησης να έχουμε πρόβλημα. Επίσης, το πρόβλημα θα έχουμε και με τη σχετική χρηματοδότηση του ΕΦΣΥ. Ε, επίσης, τι ωραία που έχουμε και την Κομισιόν εδώ. Δύο ερωτήσεις προς αυτήν. Το ελεγκτικό συνέδριο ανησυχούσε για το γεγονός ότι η χρηματοδότηση και το κλίμα δεν είχε φτάσει στο επίπεδο του 20%. Από του υπολογισμού ε, βρίσκουμε ότι αν θέλουμε να φτάσουμε στο 20% η χρηματοδότηση τα επόμενα χρόνια για το κλίμα θα πρέπει να είναι στο 22% για να φτάσουμε στο μέσο όρο του 20%. Η Κομισιόν θέλει να μου πει τι προτίθεται να κάνει για να φτάσουμε στο 20%. Και αυτή η μείωση των... της χρηματοδότησης του LIFE η πολύ απότομη αυτή μείωση, από πού προέρχεται. Ήταν πάντα πολύ αποτελεσματικό αυτό το πρόβλημα. Από πού και ω πού λοιπόν προέκυψε αυτή η απότομη μείωση τη χρηματοδότηση του LIFE. Μπορεί η Κομισιόν να μα εξηγήσει λιγάκι την αιτία. Είναι δύο συγκεκριμένε ερωτήσει προ την Κομισιόν. Εγώ σα υποστηρίζω απόλυτα, Πρόεδρε, με κάποιε επιπρόσθετες τροπολογίε όμω προ την κατεύθυνση τη δική σα ούτω ή άλλω. Ευχαριστώ, κύριε Ο κύριος ε, από το EFDT δεν είναι εδώ, κυρία Ντονάνο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την έκθεσή σας. Χαιρόμαστε που οι δημοσιονομικές υποχρεώσεις για το κλίμα φτάνουν περίπου στο 20%. Όμως, πρέπει να επιμεριστούμε τις προσπάθειες όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο αυτοί που συνεισφέρουν καθαρά. Κάθε μία από τις χώρες ε, την αφορά η κλιματική πρόκληση και επομένως θα πρέπει να εμπλακεί με χρηματοδότηση. Πέρα από το 8% των υποχρεώσεων για τη βιοπικιλότητα, πρέπει να στηρίξουμε μια, την καταπολέμηση όλων των παραγόντων που απειλούν τη βιοπικιλότητα. Ε, Παραδείγματο χάρη τα χημικά φυτοφάρμακα και κυρίως τα νεονικοτινοειδή. Ε, η παραγωγικότητα που επιβάλλει ε, η ΚΑΠ ή ας πούμε το μονοπόλιο των σπόρων είναι τεράστιο πρόβλημα. Δεν θέλουμε απλώς να αυξάνουμε συνεχώς τον προϋπολογισμό για να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα. Η αύξηση των 29 εκατομμυρίων ευρώ για το πρόγραμμα LIFE γίνεται στα πλαίσια της ε, προγραμματισμένης απώλειας της ε, καθαρής συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου μετά από τον Brexit. Αυτή η αύξηση θα σημάνει προφανώ αύξηση των συνεισφορών των άλλων κρατών μελών. Σε ό,τι αφορά τι δαπάνε για την υγεία, ε, δεν έχει κανένα νόημα προπολογισμό αν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προπομπό υιοθετώντα μια φιλόδοξη νομοθεσία, παραδείγματο χάρη για του ε, ενδοκρινικού ε, διαταράκτε ή τη γλυφοσάτη. Επίση, για την υγεία. Θα πρέπει να προσπίσουμε ε, και για τις μεταφορές. Θα πρέπει να σταματήσουμε να υποστηρίζουμε τα διασυνοριακά, τα διευρωπαϊκά δίκτυα που, που μειώνουν την ποιότητα του αέρα. Επίσης, το 0,44% υπέρ της υγείας δεν έχει τίποτα εκπληκτικό. Η προστασία και η βελτίωση της ανθρώπινης υγείας είναι αρμοδιότητες της Ένωσης που στην πραγματικότητα στηρίζουν ή συντονίζουν, συμπληρώνουν τη δράση των κρατών μελών. Ε, τα κράτη-μέλη έχουν τα περισσότερα προνόμια στην υγεία, με βάση το άρθρο 6 της ε, Συνθήκη για τη Λειτουργία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίση, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η αύξηση πάνω από 7% των υποχρεώσεων για τον μηχανισμό προστασία ε, Αστικής και πολιτική προστασία τη Ένωση καλύπτει επίγουσε ανάγκε όπω πυρκαγιές στα δάση, πυρετό έμπολα, θαλάσσια μόλυνση, σεισμοί και όλα αυτά θα τα αναφέρω στις τροπολογίες μου. Ευχαριστώ. Thank ε, Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκέρλινγκ ήρθε στο μεταξύ. Άρα μπορείτε να σχολιάσετε από πλευράς του ECR για θέματα προϋπολογισμού. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώς με αυτή την ευκαιρία επειδή είμαι σύνδεσμος με την ΕΚΑ, να σας μιλήσω για τον προϋπολογισμό. Θα διανύμω τροπολογίες για το προσωπικό για την ΕΚΑ για το 2017 να παραμείνει το προσωπικό και σε αυτό θα ήθελα να σας επισύρω την προσοχή. Τα μέλη τώρα, υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να λάβει το λόγο για θέματα προϋπολογισμού. Εάν όχι, θα ήθελα η Επιτροπή να σχολιάσει. Έχετε το λόγο. Όσο αφορά τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΤΕ, θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια ως προς το Brexit και τον προϋπολογισμό. Ε, ο προϋπολογισμός λαμβάνει υπόψη και το κόστος του Brexit και όπως ξέρετε εμείς θα υποβάλουμε έναν ε, συμπληρωματικό προϋπολογισμό σε σχέση με το συνολικό κόστος, σε σχέση με την αποκατάσταση του προϋπολογισμού μετά τις περικοπές του Συμβουλίου. Ε, μάθαμε ότι θα αποκαταστήσετε όλες τις δαπάνες όπως είχαν αρχικά προβλεφθεί. Άλλος, κάποιος άλλος. Thank you, Ευχαριστώ. Από τη Γενική Διεύθυνση της Επιτροπής από τη Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου, με συγχωρείτε. Θα ήθελα να σας μιλήσω για το κλίμα και το live. Από όσο ξέρω, ε, ήδη ε, γίνεται συνεδρίαση και αν μας επιτρέπετε θα επανέλθουμε να σχολιάσουμε το απόγευμα, αργότερα το απόγευμα. Ναι, βεβαίως μας, ε, μας ενδιαφέρουν τα σχόλιά σας, αλλά ε, φυσικά αν λήξει εγκαίρως η συζήτηση που προβλέπετε. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει μία απάντηση από πλευράς της Επιτροπής θα πρέπει να κατανοήσουμε τη θέση του Συμβουλίου. Εντάξει. Σας ευχαριστούμε πολύ για τις ε, παρατηρήσεις. Βλέπω ευρεία συνένεση επί του θέματος. Όλα όσα ελέγχθησαν λογικά και έχετε χρόνο να υποβάλλετε και τροπολογίες και θα ήθελα οι σύνδεσμοι με τους οργανισμούς να υποβάλουν τροπολογίες σε σχέση με τις ε, περικοπές και τον προϋπολογισμό των οργανισμών. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι στις 12 Ιουλίου στις 11 είναι η προθεσμία για τις ε, τροπολογίες και όπως σας είπα αναμένουμε τη θέση του Συμβουλίου μεταξύ 20 και 24 Ιουλίου. Και τότε θα υποβάλω τροπολογίες αν γίνουν περικοπές για την αποκατάσταση των εγγραφών μέχρι το τέλος του Ιουλίου και θα ψηφίσουμε για αυτή τη γνωμοδότηση στις 31 Αυγούστου που θα είναι η πρώτη μέρα εργασίας μετά το καλοκαίρι. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να έχω απαντήσεις από την Επιτροπή. Ας προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, που είναι οι ανταλλαγές απόψεων με τον κύριο Γκέρ Ντάνσετ. Σας καλωσορίζουμε. Ξέρετε τον κύριο Ντάνσετ, εκτελεστικό διευθυντή της ΕΚΑ. Πρόκειται για την ετήσια ανταλλαγή απόψεων με στα πλαίσια του τακτικού διαλόγου μεταξύ του Οργανισμού και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα έχουμε την δυνατότητα να συζητήσουμε το πρόγραμμα εργασίας, ιδιαίτερα του στρατηγικού στόχου μέχρι το 2018 ε, σε σχέση με την μεγιστοποίηση της διαθεσιμότητας της ε, πληροφορίας υψηλής ποιότητας, συνεργασία με τις εθνικές αρχές και τους εμπλεκόμενους φορείς σε σχέση με τις χημικές ουσίες, καθώς και η αντιμετώπιση του νομοθετικού έργου αποτελεσματικά, με βάση και τις περικοπές. Σε σχέση με την ειδική νομοθεσία, δυνάμει της ΕΚΑ, ο εκτελεστικός διευθυντής θα μας μιλήσει για την εφαρμογή του κανονισμού ε, REACH και για τα μελλοντικά προγράμματα. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για τις συνέπειες του προσχεδίου προϋπολογισμού για το 2018 για τον οργασμό. Ξέρω ότι αυτοχρηματοδοτήστε εν μέρη και φυσικά οι ευρωπαϊκές βιομηχανίες επιδοτούνται και από τον κοινοτικό προϋπολογισμό, όπως είπα και στην παρουσίαση του προϋπολογισμού, Μιλάμε για ένα γενικότερο σχέδιο ως προς τις δαπάνες προσωπικού. Δεν υπάρχει ειδικό προσωπικό, επιπρόσθετο προσωπικό για τους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες και επειδή υπάρχουν συγκεκριμένες κυρώσεις για την ε, μη ολοκληρωτική χρήση του προϋπολογισμού 16 θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ζήτημα της περιορισμένης χρήσης των κονδύλιων του προϋπολογισμού. Σας δίνουμε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για τα θέματα που αναφέρατε, ελπίζω να επανέλθω στο τμήμα ερωτήσεων και απαντήσεων. Έχω ετοιμάσει και μια παρουσίαση, την οποία θα ήθελα να διαβάσω, που καλύπτει εν μέρη τα στοιχεία τα οποία με ρωτήσατε. Κυρία Πρόεδρε, Αντιπρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτέ, με μεγάλη χαρά εμφανίζομαι μπροστά σα και έχω την ευκαιρία αυτή νωρίτερα από ό,τι συνήθω ε, να σα σας μιλήσω. Τελειώνει η δεκαετής ε, περίοδος ε, της θητείας μου και θέλω να σκεφτούμε λιγάκι τι σήμαινε αυτή η δεκαετία ε, για μένα προσωπικά καθώς και την Ευρωπαϊκή Ένωση και περιμένω να ακούσω βεβαίως τις ερωτήσεις και να σας απαντήσω. Όταν κοιτάμε το παρελθόν, ε, μερικές φορές ο χρόνος μας παίζει παιχνίδια. Ε, μερικά πράγματα μοιάζουν πολύ πρόσφατα ε, και παράλληλα ε, μια ολόκληρη ζωή έχει περάσει. Έτσι αισθάνομαι και εγώ. 2007. Δέκα χρόνια που πέρασαν πολύ γρήγορα. Α σα θυμίζω κάποια, κάποια έτσι βασικά στοιχεία για να σα ε, φρεσκάρω τη μνήμη. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία ε, μπήκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νέα κράτη-μέλη μπήκαν στο Σέγγεν. Το διακυβερνητικό πάνελ για την κλιματική αλλαγή είπε ότι η αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη είναι ανθρωπογενής. Και τα πρώτα σημάδια τη παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση εμφανίστηκαν όταν κατέρευσε η Lehman Brothers και η PNP Paribas ε, δεν επέτρεψε την την απόσυρση ε, χρημάτων. Ε, αυτά ήταν κοσμεστικά γεγονότα. Ε, παράλληλα, στο δεύτερο πάτωμα ενό μεγάλου κτηρίου ε, στο κέντρο του Ελσίνκη, εγώ και δέκα συνάδελφοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκινήσαμε να στείλουμε την ε, υπηρεσία την ΕΚΑ. Ήταν πολύ έντονε αυτέ οι πρώτε μέρε. Ε, ένα χρόνο μετά τέθηκε σε ισχύ το ΡΙΚΣ. Όλοι ενδιαφερόμαστε από αυτέ τι προκλήσει. Ε, το να μπορέσουμε πούμε, να επιτρέψουμε στις επιχειρήσει να προκαταχωρήσουν ε, χημικές ουσίες μέσα στην προθεσμία τη 1 η Δεκεμβρίου του 2008. Δεκάδες χιλιάδε επιχειρήσεις ουσιαστικά καταχώρησαν ε, τις χημικές ουσίε, 20 φορές περισσότερες από ό,τι περιμέναμε. Ε, όσοι από εσά έχουν ξεκινήσει οτιδήποτε από το μηδέν θα καταλαβαίνετε πόσο αγωνιώδης ήταν αυτή η στιγμή. Ε, να σας πω λοιπόν δύο πράγματα για μένα. Εγώ άρχισα να δουλεύω τον Ιανουάριο του 2007 ως ε, προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της υπηρεσίας και μετά ε, πήρα αυτή τη θέση ε, στα πλαίσια της πρώτης ε, θητείας μου. Θα θυμάστε ότι δεν ήταν όλοι υπέρ αυτού του διορισμού. Ήμουν η υπάλληλο τη Κομισιόν, πρώην τμήματάρχη ε, του τμήματο Rich DG Enterprise και πολλοί από εσά και πρώην συνάδελφοί σα ε, ανησυχούσαν ότι θα είμαι πολύ υπέρ τη Κομισιόν και πολύ θα εστιάζω πολύ ε, στο θέμα των, ε, της βιομηχανίας. Δυσκολεύτηκα πάρα πολύ, ειδικά στην πρώτη ακρόαση σε αυτό το κτίριο. Ε, να καταλάβω, έπρεπε να καταλάβω τις ανησυχίες ε, και να δικαιολογήσω την εμπιστοσύνη που μου δείξατε και να ξεπεράσω τα όρια της ε, εμπειρίας μου. Ε, χρειάστηκε να ασχοληθώ ε, με πολλά θέματα, με τις ανησυχίες των stakeholders. όταν είσαι επικεφαλής μια τέτοια ε, υπηρεσία, καταλαβαίνει ότι ο ρεαλισμό, η ταπεινοφροσύνη, η διαφάνεια και η τιμιότητα είναι σημαντικά ε, μαζί με την ε, επίγνωση ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο. Στην περίπτωση του ΕΚΑ ε, έπρεπε ο κόσμο να συνεργαστεί. Ε, Χωρί τη συνεργασία των επιχειρήσεων, χωρί τη συνεργασία των κρατών μελών, τα οποία θα μα διέθεταν του εμπειρογνωμονέ του, χωρί τι αρχέ ε, εφαρμογή να κάνουν αυτό που έπρεπε, χωρί υπηρεσίε τη Κομισιόν, να φτάνουν σε κοινέ θέσει, χωρί την ε, συμμετοχή των stakeholders, χωρί τι προκλήσει που μα έθεταν, χωρί ε, την ε, δέσμευση και το ζήλο του προσωπικού μα, δεν θα ήμασταν σε θέση να πούμε σήμερα κάποια θετικά πράγματα όπω αυτά που σας, θα σα πω. Πρέπει να αναγνωρίσω και να ευχαριστήσω επίση την πόλη του Ελσίνκη που, ε, ήταν η, που μα υποδέχτηκαν Καθώ και το φιλανδικό κράτο. Ε, φοβερή ήταν η υποστήριξή τους ε, με το κατάλληλο κτίριο. Ε, υπήρχε η υπογεγραμμένη συμφωνία για την έδρα, το νομικό καθεστώ για το προσωπικό, ε, ευρωπαϊκό σχολείο για τα παιδιά μα. ήταν και εξακολουθούν να είναι μοντέλο αποτελεσματικότητας και θερμής υποδοχής από πλευράς ενό μιας χώρας που υποδέχεται μια τέτοια υπηρεσία. Ε, εξακολουθώ να είμαι, είμαι πάρα πολύ υπερήφανος που έπαιξα το ρόλο μου ε, στο τιμόνι της ΕΚΑ και κατάφερα ε, αυτός ο οργανισμός να είναι ανοιχτός ε, και επίσης θα κάνω ό,τι μπορώ ούτως ώστε να παραδώσω στον διάδοχό μου μια υπηρεσία η οποία είναι στο ύψος των αξιών της. να είναι ανεξάρτητη, να εμπνέει εμπιστοσύνη, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και να προωθεί την ευημερία. Ε, επίσης, ε, θα, τη θα ένα πολύ καλό προσωπικό που θέλει να προστατεύσει την ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον και δέχεται κάθε πρόκληση. Ε, η ΕΚΑ ε, κάνει ό,τι μπορεί για την Ευρωπαίο πολίτη αλλά και για τις επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν ένα τεράστιο καθήκο, μια τεράστια πρόκληση το να με το REACH, το BPR, το CLP και το PICA. Δέκα χρόνια μετέτρεψαν, άλλαξαν τελείω τη ζωή μου. Ε, με πίεσαν με κάθε τρόπο. Ε, μου έδωσαν μια τεράστια ευκαιρία όλα αυτά, ως καταλαβαίνετε ότι βεβαίω η δουλειά τη ΕΚΑ δεν σταματάει με την αποχώρησή μου. Σε λίγου μήνε κάποιο άλλο θα είναι στο τιμόν τη ΕΚΑ ε, και θα σας θα έρθει εδώ να, παρουσιάσει, να παρουσιαστεί όπως έκανα εγώ 10 χρόνια πριν ε, και θα ελπίζει να, το, να εγκρίνεται το διορισμό του. Όποιο και αν είναι, αυτό ή αυτή θα χρειαστεί την υποστήριξή σα. Ε, θα αντιμετωπίσει πολλέ προκλήσει, μερικέ από αυτέ ε, σαν τι δικέ μου, αλλά και πολλέ καινούριε. Μία διαρκή πρόκληση είναι να έχει τα λεφτά και το προσωπικό του ώστε να κάνει το έκατε δουλειά σωστά. Κάθε οργάνωση το αντιμετωπίζει, αλλά πολύ περισσότερο η ΕΚΑ, όπου πολύ περισσότερη δουλειά και όλο και περισσότερε απαιτήσει από του stakeholders ε, μας βαραίνουν ε, με λιγότερου πόλου. Ε, είχα εμπειρία από πρώτο χέρι για τι απαιτήσει που υπάρχουν εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση όταν επισκεφθήκα την Κίνα πρόσφατα. Οι Κινέζοι θέλουν να σεβαστούν το REACH, ε, οι εξαγωγεί του το χρειάζονται και έχουν μια τάση προ μεγαλύτερη ε, περιβαλλοντική προστασία και προστασία τη υγεία. υγεία. Είναι στο συμφέρον τη Ευρώπη να του βοηθήσει να συμμορφωθούν. Ασφαλίστερα προϊόντα από την Κίνα είναι καλό για όλου μα. Ο ε, διαδοχός μου θα χρειαστεί τη βοήθειά σας για να τετραγωνίσει τον κύκλο. Ε, το ΕΚΑ έχει ένα τεράστιο σώμα πραγματογνωμοσύνης. Πρέπει να το αξιοποιήσουμε αλλά, και πρέπει να κάνουμε περισσότερα, αλλά θα πρέπει ο διάδοχός μου να έχει και το προσωπικό και τα λεφτά για να το καταφέρει. Ε, να σας ρωτήσω το εξή. Γιατί τα θεσμικά όργανα χρειάζονται τέτοιο αυστηρό έλεγχο πάνω ε, στο προσωπικό των οργανισμών, ειδικά όσων εισπράττουν ε, τέλη και έχουν τη δυνατότητα να αυτοχρηματοδοτηθούν. Ε, ποιοι είναι οι κίνδυνοι που περιορίζεται με τον έλεγχο αυτών. Και επιπλέον, ε, αξίζει τον κόπο κάθε χρόνο να δίνεται αυτή η μάχη με την Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, για του αριθμού των έκτακτων υπαλλήλων, με βάση τα νούμερα των τελευταίων 10 χρόνια θα έλεγα ότι οι όριμοι ε, οργανισμοί που θα πάνε καλά θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να αυτοδιαχειρίζονται τι υποθέσει του και να έχουν και τον προπολογισμό. Και βεβαίω θα πρέπει να λογοδοτούν σε εσά για αυτά που κάνουν. Μία άλλη πρόκληση πολύ βασική που παραμένει και θα την ο διάδοχός μου είναι η ποιότητα των δομένων που παρέχουν οι εταιρείε. Ο REACH έχει δημιουργήσει υψηλέ απαιτήσει στις εταιρείε για να παρέχουν δεδομένα για τις ε, ουσίες που παρασκευάζουν, χρησιμοποιούν και ε, πολλούν και πρέπει να πούμε ότι η ποιότητα των δεδομένων δεν είναι πάντα υψηλή. Φυσικά και υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, Όμω, εάν τα δεδομένα για μια ουσία δεν συμμορφώνονται, αυτό επηρεάζει την ικανότητά μας να εντοπίσουμε επικίνδυνε ουσίε και να διαχειριστούμε τους κινδύνους που αυτές ε, θα ε, δημιουργήσουν. Και η αντιμετώπιση λοιπόν του θέματος των ατελών δεδομένων είναι μια πρόκληση που θα συνεχίσουμε να έχουμε για να επιτύχουμε τους στόχους του ΡΙΤΣ. Γι' αυτό λοιπόν έχω πιέσει για να δημιουργηθεί μια τομεακή συνεργατική προσέγγιση όπου ε, θα ε, υπάρχει κοινή ευθύνη από όλους ε, έτσι ώστε να επικαιροποιούν τα χαρτοφυλάκια τους. Η τρίτη πρόκληση που θα αντιμετωπίσουμε είναι μία που γνωρίζετε πολύ καλά, να έχουμε δηλαδή αρκετές πληροφορίες για, τους, ε, για τα μη τυπικά είδη ή ε, μορφές από ουσίες όπως των ενδοκρινικών διαταρακτών, των πολυμερών και τα ανανοηλικά. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας για να συλλέξουμε τα δεδομένα για τις ε, ε, πολύ μικρές για τις νάνομορφές των ουσιών και όπως ε, ανέφερα πρέπει τα δεδομένα να είναι αξιόπιστα έτσι ώστε να μπορούμε και εμείς να αξιολογήσουμε τον κίνδυνο που ε, αυτά αποτελούν για τους ανθρώπους και το περιβάλλον και θεωρώ πως κάποια στιγμή Ελπίζω ε, πως θα φτάσει η στιγμή που η Κομισιόν θα έχει το θάρρος ε, να ε, κλείσει αυτό το κενό που υπάρχει στις νανοουσίες και η ΕΚΑ θα αποκτήσει ισχυρότερη εντολή για να αντιμετωπίσει τις εταιρείε που δεν συμμορφώνονται. Και ελπίζω να δείτε και εσείς την πρώτη φάση του νανοπαρατηρητηρίου, την οποία ξεκινήσαμε στις 14 Ιουνίου. Είναι μια καλή αρχή και προσπαθεί να συλλέξει υλικό από διάφορες πηγές για να δημιουργήσει δημιουργήσει μια αντικειμενική βάση δεδομένων για τα ανανοηλικά. Και το περιεχόμενο του παρατηρητηρίου ε, θα διευρυνθεί, θα αυξηθεί με τον καιρό και ελπίζω να συνεισφέρει σημαντικά στην ε, συζήτηση για τα ανανοηλικά και τον αντίκτυπό του. Οι ευκαιρίε τώρα που έχουμε για το μέλλον ε, θα είναι επίσης πάρα πολλές. Έχουμε ε, τους ε, παγκόσμιους στόχους για τη βιωσιμότητα το 2030, τις πολιτικές για την οικονομία, μη τοξικό περιβάλλον, ε, ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ηθικές επενδύσεις, προστασία εργαζομένων και καταναλωτών, κλιματική αλλαγή και την καταπολέμηση της ρήπανσης από πλαστικά. Όλα αυτά για να τα αντιμετωπίσουμε πρέπει να κατανοήσουμε καλύτερα τη σύνθεση των προϊόντων και να μειώσουμε την έκθεση σε ουσίες που είναι βλαβερές για τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Οι καταναλωτές απαιτούν πιο ασφαλή, πιο ε, ηθικά ε, προϊόντα τα οποία θα έχουν, ε, θα είναι προϊόντα τα οποία δεν θα βλάπτουν τους χρήστες κατά τη διάρκεια της χρήσης τους. Και οι νομοθέτες, οι καταναλωτές και οι επιχειρηματίες πρέπει να βρίσκονται σε και να έχουν κοινή άποψη έτσι ώστε να γίνει κάτι θετικό. Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για την ΕΚΑ είναι να συγκεντρώσει τα δεδομένα και την εμπειρογνωμοσύνη που συνέλεξε ο ΡΙΤΣ για να στηρίξει αυτές τις εξελίξεις. Και πρόσφατα ε, καταφέραμε να δημιουργήσουμε την πρώτη βάση δεδομένων ε, του ΡΙΤΣ που μπορούν να κατεβάσουν ε, διαδικτυακά οι ερευνητές θα γίνουν κι άλλα στο μέλλον. Θα υπάρχει ανταλλαγή δεδομένων, θα υπάρχουν αλγόριθμοι, συλλογή δεδομένων, έτσι ώστε τα ε, δεδομένα στο REACH να δίνουν περισσότερη αξία στον πολίτη και να στηρίζουν και τις πολιτικές μας. Αυτό μπορούμε να το καταφέρουμε χτίζοντας πάνω στις επενδύσεις που έχουν ήδη γίνει συλλογικά και ε, να μην ξεχάσω να αναφέρω το σχεδόν ένα δισεκατομμύριο ευρώ που έχει δαπανηθεί ε, για την ΕΚΑ τα τελευταία 10 ε, χρόνια. Το, το 60% του ποσού αυτού να πω επίσης ότι έχει καταβληθεί με τη μορφή τελών από επιχειρήσεις. Η επόμενη ευκαιρία είναι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, με το να τους δίνουμε εύκολη πρόσβαση στα δεδομένα για να ε, παράγουν πιο ε, ασφαλή χημικά. Και κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να ε, προσφέρω, να εκτελέσω το καθήκοντά μου τα τελευταία δέκα χρόνια. Ελπίζω να σας έπεισα ότι ήμουν ο κατάλληλος άνθρωπος ε, για αυτήν την θέση και θα ήθελα επίσης ε, να δείξω την ευγνωμοσύνη μου και για την δουλειά που έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές που λειτουργούν ως σύνδεσμοι μεταξύ ημών και ημών, η Σάτου Χάση και η Τζούντι Γκέρλινγκ. Είναι άτομα που έχουν συνεχιζόμενη αναλαμβάνει δέσμευση και έχουν κάνει υποδειγματική δουλειά. Στην αρχή της θητείας μου δημιουργήσαμε μια εταιρική ταυτότητα, δημιουργήσαμε ένα όρομα και μια αποστολή, αξίες που ε, μας συνόδευαν σε όλη τη διάρκεια της ε, θητείας μου. Η ΕΚΑ στόχο έχει να είναι η μεγαλύτερη ρυθμιστική αρχή παγκοσμίω για την ασφάλεια των ε, χημικών και νομίζω πως ε, χωρίς να είμαι υπερβολικά αισιόδοξο, ότι Έχουμε ε, καταφέρει πολλά προς αυτό. Έχουμε σχεδόν επιτύχει αυτό και νομίζω πως μπορώ να αποσυρθώ από την θέση μου γνωρίζοντας ότι έχω κάνει ό,τι μπορώ για να μας φτάσω σε αυτό το σημείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα τώρα να ακούσω με χαρά τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ ενδιαφέρον από τους συναδέλφους να προβούμε σε ένα διάλογο. Έχω έναν κατάλογο μπροστά μου αλλά η κυρία Γκέρλινγκ έχει καταρχήν το λόγο που είναι και ο σύνδεσμος με τον οργανισμό σας. Κυρία Γκέρλινγκ, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ και σας ευχαριστώ και για την ομιλία σας που ήταν κάπως διαφορετική από το ε, σύνηθες ως ε, αποχαιρετιστήρια ομιλία. Θα ήθελα λοιπόν να υποβάλω αρκετές ερωτήσεις, λίγο διαφορετικές από τις συνηθισμένες Έχετε ταξιδέψει στην Κίνα πρόσφατα, από ό,τι μας ε, είπατε. Θα μπορούσατε να μας πείτε ορισμένες σκέψεις ε, για τη θέση του ΡΙΤΣ ε, μέσα στα πλαίσια του παγκοσμίου ρυθμιστικού πλαισίου, γιατί υπάρχει μία, θα μπορούσα να πω, ε, ανάλυση του ότι το ΡΙΤΣ είναι πολύ ανταγωνιστικό σε σχέση με το αντίστοιχο πρόγραμμα τον είπα. Και επειδή ο κύριος Τραμπ είναι πολύ απασχολημένος, και δεν ενδιαφέρεται τόσο για τα κλιματικά, δεν ξέρω ποια είναι η θέση του ε, για τα χημικά και δεν ξέρω κατά πόσο το δικό του πρόγραμμα αντιστοίχως είναι εξίσου εύρωστο. Γιατί ξέρουμε γιατί ξέρουμε ότι οι ΙΠΑ ήθελαν η Κίνα να εγκρίνει το δικό τους πρόγραμμα. Δεν ξέρω κατά πόσο υπάρχει αυτή η θέση. Ως προς την προθεσμία του 2018 για τις ΜΜΕ, ξέρω ότι έχετε καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για να ε, βελτιώσετε τα πράγματα για τις ΜΜΕ και επειδή θα φύγετε πέντε μήνες νωρίτερα από το προβλεπόμενο, δεν ξέρω πώς ε, βρίσκεται ότι μπορεί να τηρηθεί αυτή η προθεσμία για τις ΜΜΕ. Θα κάνουμε ένα γύρο ερωτήσεων και μετά θα απαντήσετε. Ευχαριστώ πολύ. Τι να πω και εγώ η ΕΚΟ δεν θα είναι ίδια, λέει ο κύριος Πόκ. Και θα ήθελα να ασχοληθούμε με επιμέρους σοβαρά ζητήματα όταν δούμε τις ε, χημικές ουσίες και τα βιοκτώνα και πώς αποτιμώνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση Έχω και την προσωπική μου άποψη ότι ίσως υπάρχουν κενά και θα ήθελα τις δικές σας απόψεις όταν αξιολογούμε την επικινδυνότητα των βιοκτώνων ή των φυτοκτώνων πολλές φορές δεν βλέπουμε τις παρενέργειες αυτών των χημικών και έχω Έχω και τη γλυφοσάτη που είναι μια ένωση που με απασχολεί ιδιαίτερα, είναι αγαπημένη μου και νομίζω ότι τη γνωρίζετε. Ε, πρόκειται για ένα αντιβιωτικό που χρησιμοποιείται. Και τι κάνουμε, στην ουσία ψεκάζουμε τις καλλιέργειες με αυτό το αντιβιωτικό χωρίς να γνωρίζουμε επακριβώς τις παρενέργειες, δηλαδή κατά πόσο θα μπορούσε να έχει ε, συγκεκριμένες αρνητικές συνέπειες, ιδιαίτερα σε, ως προς την ε, γενικότερη μεταχείριση αυτής της ουσίας. Με τη δεκαετή σας πείρα, με βάση αυτή τη δεκαετή σας πείρα, πόσο μακρόπνοα θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την νομοθεσία μας εάν υπάρχουν κίνδυνοι και από πλευράς ε, μεγάλων επιχειρήσεων και πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Φλόρενς. Μάλιστα, κύριε Τάνσεν. Δεν ήθελα αρχικά να τοποθετηθώ πάνω στο θέμα αυτό. Θα ήθελα όμως να σας υπενθυμίσω ότι πολλά χρόνια πριν, όταν ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Περιβάλλοντος, είχαμε επεξεργαστεί όλη τη δεσμή μέτρων για τον κανονισμό REACH. Ήταν περίπου χίλιες σελίδες, μεγάλος όγκος. Και όταν άρχισε η συζήτηση λοιπόν στην αρχή δεν ξέραμε πώς ε, να προχωρήσουμε, δεν ξέραμε πώς να σηκώσουμε αυτό το αεροπλάνο στον αέρα. Τεράστια ο όγκος δουλειάς. Όμως, ε, επίσης δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημά μας. Δεν υπήρχε πουθενά στον κόσμο κάποια παρόμοια περίπτωση. Ένα παράδειγμα, κάτι να μπορούμε να βασιστούμε πάνω του. Ε, ευτυχώς όμως, το καταφέραμε χωρίς όμως ε, παράπλευρες απώλειες. Μάλιστα με κατηγόρησαν στην πατρίδα μου ότι ο Φλόρενς διέλυσε την γερμανική βιομηχανία. Ακούσαμε πάρα πολλά αρνητικά όμως ε, το γεγονός είναι ότι μόνο τα αρνητικά ακούγονται πολύ. Μόνο 30 ή 40 προϊόντα είναι αυτά τα οποία έχουν δημιουργήσει πρόβλημα. Δεν έχουμε αξιολογήσει όμως μόνο 30-40 προϊόντα. Έργο μας είναι να ξεδιαλέξουμε από χιλιάδες προϊόντα αυτά τα 30-40, να τα εντοπίσουμε. Κύριε Ντάντσεν, νομίζω πως εσείς ε, ήσασταν πάρα πολύ τυχερός. Διότι στην αρχή του όλου εγχειρήματο ζητήσαμε βοήθεια. Δεν ξέραμε τι να κάνουμε, δεν ξέραμε πώς θα καταφέρουμε να δημιουργήσουμε όλες τις αναγκαίες συνδέσεις, όλες τις γέφυρες για να συνδεθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τις ε, δομές μας. Δεν ξέραμε τι θα κάνουμε και πώς θα το κάναμε. Εσείς όμως σίγουρα βοηθήσατε πάρα πολύ τη βιομηχανία της επιχειρήσης. Όμως, κύριε Ντάνσεν, να κάνω και ένα αστείο. Εάν επιτραπεί να κλωνοποιήσουμε ευρωϊπαλλήλους, να είστε σίγουρος πως εσείς θα είστε ο πρώτος που θα κλωνοποιηθεί. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ντονάνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Διευθυντή. Πρώτη ερώτηση. Αφορά την εφαρμογή του καονισμού REACH και την περιπλοκότητα των διαδικασιών αξιολόγησης των κινδύνων από τις επιχειρήσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει κάτι το άσχημο εδώ. Μερικές δηλαδή ε, επιχειρήσεις προσπαθούν να επιλέξουν ε, πιο περίπλοκα προϊόντα λιγότερα περίπλοκα προϊόντα ή να πάνε προς προϊόντα που δεν χρειάζεται καταχώρηση. Τι μέσα έχετε ούτως ώστε να μην τους επιτρέψετε κάτι τέτοιο. Δεύτερον, τη διαχείριση του προσωπικού στο εσωτερικό της ΕΚΑ. Ξέρω ότι πρέπει να σέβεστε κάποιους στόχους πολύ συγκεκριμένους ε, για τη μείωση του προσωπικού, Φερρυπίν. Όμως δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση για να καλυφθούν τα θέματα ε, των ενδοκρινικών διαταρακτών. Τελικά, τι θα κάνετε ακριβώς με αυτό το θέμα. Ε, πώς θα μπορέσετε να καλύψετε αυτές τις ανάγκες και να υπάρξει άτομο το οποίο θα ασχοληθεί με τους ενδοκρινικούς διαταράχτες. Θα επιλέξετε δηλαδή ανάμεσα σε κάποια θέματα. Ε, κυρία ε, Γκέρλιν, ε, ευχαριστώ κύριε. Ευχαριστώ κυρία, κυρία Ντάνσετ. Περάσατε 10 χρόνια ε, και ετοιμάστε να πάρετε σύνταξη. Ε, μπορείτε να δείτε λοιπόν τα πράγματα αντικειμενικά, τις προκλήσεις που μας ε, περιμένουν κτλ. Αυτά που κατάλαβα από την παρουσίασή σας και κάτι που θα ήθελα να σας ρωτήσω, αντί να εστιάσουμε στο παρελθόν, είναι να σας ε, ρωτήσω ότι αυτό που μας παρουσιάζεται είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, ε, αν μου επιτρέπετε το θέτω έτσι. Ε, είπατε ότι οι κατανοτές θέλουν καλύτερα προϊόντα και πιο ασφαλέστερα προϊόντα και προϊόντα που δεν προκαλούν βλάβη στην υγεία τους και το περιβάλλον τους. Όμως, αναφέρεται και δύο προκλήσεις. Ότι ας πούμε τα δεδομένα για τις διάφορες ουσίες δεν είναι αρκετά καλής ποιότητας και αυτό επηρεάζει την ανάλυση της υπηρεσίας σας και τον εντοπισμό των κινδύνων. Και επίση είναι πάρα πολύ δύσκολο να λάβουμε πληροφορίες γιατί δεν είναι πάντα αξιόπιστες. Ε, και επιπλέον είναι κοντόθωρες ε, οι επιχειρήσεις μερικές φορές και δίνουν τα ελάχιστα δεδομένα που απαιτούνται. Αυτός ο φαύλος κύκλος πώς μπορεί να σπάσει, κατά τη γνώμη σας. Ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι η ΕΚΑ εξαρτάται από έσοδα της ίδιας της βιομηχανίας, που θα εισπράξει από τη βιομηχανία τι μέτρα μπορούν να προωθηθούν, ούτως ώστε να είμαστε σίγουροι ότι η βιομηχανία δίνει αξιόπιστες πληροφορίες, σας δίνουν δεδομένα τα οποία δεν είναι τα ελάχιστα και σας δίνει πληροφορίες που πραγματικά μπορούν να υλοποιήσουν τους στόχους της υπηρεσίας σας. Δηλαδή, ασφαλή προϊόντα για τον κόσμο, αλλά και για το περιβάλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμότατα για την παρουσίασή σας. Ήταν, όπως είπε και ο συνάδελφος Φλόρνης, λίγο διαφορετική από αυτή που έχουμε συνηθίσει. Ε, και είδα αρκετό θάρρος, αρκετή αισιοδοξία στην ε, ομιλία σας και πραγματικά μου αφήσατε την εντύπωση ότι πράγματι έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε κάτι πάρα πολύ καλό. Ε, έχω όμως κάποιους φόβους για το μέλλον. Δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον. Συζητήσαμε για τον προϋπολογισμό και μας είπατε και εσείς πως στο νέο προϋπολογισμό υπάρχει μείωση κατά δύο θέσεις του προσωπικού. Βλέπουμε ότι και ε, για, για τον ΕΦΣΑ υπάρχει η ίδια Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο, ιδιαίτερα με τόσα χημικά που ε, εμφανίζονται στην αγορά. Ε, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει αύξηση. Ταυτόχρονα βλέπουμε πως αυξάνεται ο όγκος δουλειάς, μειώνεται το προσωπικό. Δεν βλέπω σωστά επιχειρήματα υπέρ αυτής της απόφασης και νομίζω ότι είναι λάθος. Και ε, επιτρέψτε μου και μια έτσι ρητορική ερώτηση. Θα υπάρξουν στο μέλλον περισσότερα χημικά, θα έχει ο ΕΚΑ περισσότερη δουλειά. Αυτό τι θα σημαίνει. Θα σημαίνει πως ε, εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε σε θέση να διαθέσουμε περισσότερους πόρους για να κάνετε σωστά τη δουλειά σας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπράνεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Διευθυντά, που ήρθατε εδώ. Αναφέρατε ότι ο ΕΚΑ έχει την έδρα στην Φιλανδία. Η Φιλανδία είναι μια χώρα η οποία φιλοξένησε εξαιρετικά τον οργανισμό αυτόν. Εγώ είμαι Βρετανός, Ευρωβουλευτής και όπως γνωρίζετε η Βρετανία θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν αρκετοί οργανισμοί με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τους οποίους θα χάσουμε. Και δεν θέλω τώρα να σας ζητήσω να τοποθετηθείτε πολιτικά, αλλά να σκεγγραφίσετε κατά τη δική σας άποψη, ως επικεφαλής ενός τέτοιου οργανισμού, ποια ήταν τα ωφέλη για τη Φιλανδία του να φιλοξενεί έναν μεγάλο ευρωπαϊκό οργανισμό στο έδαφος της. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Εδώ ολοκληρώθηκαν και οι ερωτήσεις των Ευρωβουλευτών. Κύριε Ντάνσετ, θα σας δώσω το λόγο ή να δώσω πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα θέλατε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τη σειρά ως προς την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Κίνα, αυτή ήταν και η πρώτη ερώτηση, η κινέζικη κυβέρνηση ανησυχεί ιδιαίτερα με θέματα ανθρώπινης υγείας και περιβάλλοντος και θέλουμε να, έχουμε καλύτε, θέλουμε να έχουν καλύτερη νομοθεσία προστασίας των πολιτών γιατί έχουν δώσει προτεραιότητα ώστε να μην γίνονται άλλες εκρήξεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπως έγινε δύο χρόνια πριν όπου έγινε μια μεγάλη έκρηξη σε ένα χημικό εργοστάσιο και όπου σκοτώθηκαν πολλοί άνθρωποι. Προσπαθούν λοιπόν να αναθεωρήσουν το πλαίσιο και γι' αυτό η Κίνα επιδεικνύει ανοιχτό πνεύμα και αυτό το είδα σε επίπεδο διαφόρων υπουργείων για να μάθουν από μας από την Ευρώπη και για να φτάσουν σε παρόμοια επίπεδα προστασίας. Επίσης, Φαίνεται ότι θα, σε, θα πέναμε σε έναν ανταγωνισμό με την αναθεωρημένη Τόσκα, αλλά η Κίνα δεν είναι πλέον πεπισμένη ότι ο αμερικανικός τρόπος προστασίας είναι ο καλύτερος τρόπος προστασίας. Και αυτό ήταν μια μεγάλη ανακούφιση για εμάς, γιατί είχα ακούσει το αντίθετο πριν φύγω. Άρα η Ευρώπη έχει μια μεγάλη ευκαιρία να πουλήσει το δικό της πρότυπο που θα βοηθήσει στην προστασία των πολιτών στην Κίνα και επειδή η Κίνα κάνει τεράστιες εξαγωγές σε μας, έχει μεγάλη σημασία να δούμε και αυτό το σκέλος εγώ συζήτησα στο Κουανζού και στην Καντόνα. Το 75% των ε, παιχνιδιών ε, παράγονται στην Κίνα και 50% παράγεται σε μία μόνο επαρχία. Εάν λοιπόν συμβαδίζουν με τη δική μας νομοθεσία μακροχρόνια θα ήμασταν όλοι πολύ πιο προστατευμένοι. Οι τοπικές αρχές λοιπόν ήταν πρόθυμες να ανοίξουν και ένα help desk για τις επιχειρήσεις σε επίπεδο περιφέρειας και σε σχέση με τα πρότυπα και ιδιαίτερα τα μελλοντικά πρότυπα. Αυτό είναι ένα πολλά υποσχόμενο πλαίσιο. Ως προς την προθεσμία για το 2018 είναι ύψης της σημασίας, πράγματι, τα πρώτα μηνύματα δεν είναι και τόσο καλά, γιατί έχουμε λιγότερες ε, εγγραφές ε, από τις ΜΜΕ, ιδιαίτερα για τη χαμηλότερη κατηγορία. Ε, οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη λοιπόν αντιδρούν. Επίσης υπάρχουν πολλές διαμάχες για την επίδοση πληροφοριών, διότι υπάρχει και το θέμα της επιστολής πρόσβασης. Γι' αυτό τα Μητρώα ζητούν ε, δυσθεώρητες τιμές παρά το, την, πράξη, την εκτελεστική πράξη της Κομισιόν. Άρα σε επίπεδο διευθυντών στην ομάδα συνεργασίας με την Κομισιόν και τις βασικές βιομηχανικές ενώσεις το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο θα έχουμε καλύτερες κατευθυντήριες γραμμές για την τιμολόγηση ε, μίας επιστολής πρόσβασης για υψηλά επίπεδα ε, ΝΑΣ. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την πρόσβαση στην αγορά. Έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. Επίσης, ίσως υπάρχουν κίνδυνοι η τιμολόγηση αυτή του 18 να είναι υπερτιμημένη και για πρώτη φορά θα είχαμε χαμηλότερα, εισοδήμα, χαμηλότερα έσοδα από αυτά που προβλέπονταν Αρχικά είχαμε ψηλότερα, αυτό προέβλεπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τώρα φαίνεται ότι δεν θα έχουμε τόσο υψηλά έσοδα και θα είναι πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε ο οργανισμός να λάβει επιπρόσθετα κονδύλια κατά τη διάρκεια του έτους για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα όλα ζητήματα, γιατί χρειαζόμαστε τουλάχιστον 100 ε, συμβασιούχους για να μπορούν να ελέγχουν τους φακέλους και αυτό δεν γίνεται μόνο μέσω υπολογιστών. Και αυτό από μόνο του σημαίνει ότι χρειαζόμαστε 50 εργαζόμενους επιπλέον. Θα σας μιλήσω αργότερα για το προσωπικό. Το ερώτημα του κυρίου Πότς ως προς το ερώτημά του, είναι σαφές ότι υπάρχουν κενά τεχνογνωσίας που θέλουμε να κλείσουμε. Και ξέρω α, ότι ασχολείστε ιδιαίτερα με τα βιοκτώνα, τα παρασιτοκτώνα ή τις χημικές ουσίες. Σας απασχολούν ιδιαίτερα. Και γι' αυτό θα πρέπει να θέσουμε το καλό παράδειγμα για να καταγράψουμε αυτές τις χημικές ουσίες εκ των προτέρων, το συντομότερο δυνατόν, έτσι ώστε να βρεθούν εναλλακτικέ λύσεις εγκαίρως. Και αυτό αφορά και την κλειφωσάτη που μπορεί να Εμείς είμαστε υπεύθυνοι μόνο για την αποτίμηση κινδύνου. και ε, τον αναλύουμε με βάση τα κριτήρια CLP για την επικινδυνότητα. Και ε, οι επιπτώσεις ως προς τα αντιβιωτικά δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτά τα σημεία CLP και γι' αυτό δεν έχουμε νομική βάση για να μπορέσουμε να τα λάβουμε υπόψη κατά τον ε, ίδιο τρόπο. Και αυτό αφορά και τα συστατικά της γλυφοσάτης που χρησιμοποιούνται στο Roundup. Άρα δεν ξέρουμε κατά πόσο το Roundup προστατεύει τις καλλιέργειές μας. Είναι κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει μέσα στα πλαίσια της έγκρισης της γλυφοσάτης. Η ΕΦΣΑ θα αποτιμήσει τους κινδύνους περισσότερο. Και μετά φυσικά οι εθνικές αρχές θα αποφασίσουν για τα προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν για ψεκασμούς. Υπάρχει λοιπόν ε, ένας επιμερισμός ευθυνών σε αυτή τη διαδικασία. Μετά αναφερθήκατε στα έγγραφα Μονσάντο και κατά πώς θα πρέπει να αναθεωρήσουμε τον όλο τρόπο εξέτασης χημικών ουσιών, γιατί εδώ και δεκαετίες βάζουμε το βάρος των αποδείξεων της απόδειξης της επιχειρήσης. Εκείνες πρέπει να δοκιμάσουν τις χημικές ουσίες σύμφωνα με τα κριτήρια GLP και χρησιμοποιούν και ανεξάρτητα εργαστήρια. Εδώ υπάρχουν κατηγορίες και αποδείξεις ότι η Σάντο και η ΙΠΑ ε, χειραγώγησαν κατά κάποιο τρόπο ορισμένες μελέτες. Δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για χειραγώγηση των δοκιμών των εργαστηρίων με βάση αυτά που μας έχει πει η ΕΦΣΑ, αλλά εάν κινδυνεύει το σύστημά μας, θα πρέπει να ξαναδούμε τον όλο τρόπο λειτουργίας μας. Σε βάση περιπτώσει, οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να αξιολογούν καλύτερα τα αποτελέσματα των εργαστηρίων και ίσως οι βιομηχανίες θα πρέπει να πληρώνουν τις δημόσιες αρχές να κάνουν αυτές τις δοκιμές. Αυτό δεν αποτελεί τρέχουσα πρακτική και δεν μπορούμε να την αλλάξουμε μία νυχτή. Σας ευχαριστώ κύριε Φλόρενς για τα καλά σας λόγια, για το τι πέτυχα όλα αυτά τα χρόνια. Είναι γεγονός ότι όταν αρχίσαμε, όταν άρχισα εγώ με τις μελέτες αντικτύπου της ε, πρότασης προέβαλα μια συνεργατική διαδικασία έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη τις επιπτώσεις της νομοθεσίας και προσπαθήσαμε να κάνουμε δοκιμές πριν από την εφαρμογή της νομοθεσίας. Επειδή είχαμε λοιπόν αυτή τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, όχι μόνο ε, την βιομηχανία αλλά και τις ΜΚΟ και τα συνδικάτα. Προσπαθήσαμε να έχουμε μία απαιτητική νομοθεσία έτσι ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των χημικών ουσιών. Βλέπουμε ως προς το ευρωβαρόμετρο ότι έχει αυξηθεί η εμπιστοσύνη στις χημικές ουσίες την τελευταία δεκαετία και αυτό οφείλεται στο ριτς πρωτίστως. Ως προς τις ΜΜΕ είπα ήδη ότι έχουμε κάνει πολλά για να βελτιώσουμε την καθοδήγηση των ΜΜΕ, αλλά θα πρέπει η τιμολόγηση να είναι χαμηλότερη για να μπορούν να εγγραφούν στα Μητρώα. Είχα προτείνει και πιο ριζοσπαστικές λύσεις στο παρελθόν που δεν έγιναν αποδεκτές. Τώρα θα πρέπει να βρούμε λύσεις που εντάσσονται στο σημερινό νομικό πλαίσιο, έτσι ώστε να κρατήσουμε όσο περισσότερες ε, επιχειρήσεις μπορούμε στη μεγάλη αυτή βιομηχανία, γιατί εκείνες ε, αποτελούν τη μεγαλύτερη αξία για την κοινωνία. Η εφαρμογή Ο επόμενος ομιλητής μίλησε για αρνητικές επιπτώσεις. Η επόμενη με Δημήτρη ήταν στην πραγματικότητα. Εμείς έχουμε αποδείξει ότι αν υπάρχει ισορροπία ανάμεσα στην ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλον και από την άλλη την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα, αυτή είναι η σωστή ισορροπία, ούτως ώστε η νομοθεσία να έχει τις καλύτερες δυνατές ε, επιπτώσεις στο μέλλον. Με την ε, βιώσιμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της ε, βιομηχανίας, η βιομηχανία της Ευρώπης αποκτά μέλλον. Μετά, κοιτάξτε, για το προσωπικό. Ε, για πέντε χρόνια, στήσαμε μάλλον την, ε, την ΕΚΑ, πέντε χρόνια ήταν σταθερό το προσωπικό μας και μετά η μείωση. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και παρόλα αυτά κάνουμε αυτά που υποσχεθήκαμε. Ήμουν βέβαια τυχερός που αυτή η μείωση αντισταθμίστηκε γιατί δεν είχαμε μια καθαρή μείωση του προσωπικού ε, πάντως, ε, στα πλαίσια του CLP χρειάστηκε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερο προσωπικό. Είναι μια συνεχής μάχη. Και τώρα μας λένε ότι θα πρέπει να αρχίσουμε να εργαζόμαστε για τα όρια της έκθεσης ε, στο χώρο εργασίας. Ε, επίσης ε, και για τη δηλητηρίαση, ενδοκρινικούς διαταράκτες, χωρίς να έχουμε νέο προσωπικό, χωρίς να έχουμε νέους υπαλλήλους. Εμείς ξεκαθαρίσαμε ότι δεν μπορούμε να ξεκινήσουμε του χρόνου να αναλάβουμε και αυτά τα επιπλέον καθήκοντα χωρίς επιπλέον υπαλλήλους. Γιατί, όπως σας είπα, χρειαζόμαστε 100 άτομα για το Red Line, συν όλους τους επιπλέον που χρειαζόμαστε για να ελέγχουμε. Γι' αυτό ε, δεν θέλουμε οι έξι άνθρωποι που ασχολούνται με το REACH να μην μειωθούν. Αν θέλετε να το, τους μειώσετε, ας τους μειώσετε το 2019. Δηλαδή, μην, κλείσετε, μην κόψετε από τους 6 συν τους 3 που ασχολούνται με τα βιοκτώνα. Ε, γι' αυτό 6 μείον 4 ίσον 2, αυτή ήταν ε, η αρχική, ο αρχικός υπολογισμός. Στην πραγματικότητα θέλουμε όμως 6 επιπλέον άτομα. για το φαύλο κύκλο και πώς θα έχουμε από τη μία πιο ασφαλή προϊόντα, ενώ δεν έχουμε ε, όλα τα δεδομένα, πώς θα τεταγωνίσουμε αυτόν τον κύκλο. Όταν εγώ μίλησα για κοντόθωρες επιχειρήσεις, μιλούσα για τι επιχειρήσει νενοηλικών περισσότερο. Γιατί παρά το γεγονός ότι η ερμηνεία της Κομισιόν και δική μα είναι ότι το REACH καλύπτει όλες τις ουσίες στην πραγματικότητα ε, η βιομηχανία συστηματικά αμφισβητεί το γεγονός ότι καλύπτονται και τα νοηλικά από το REACH. Και από τις πρόσφατες ε, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου Προσφυγών ε, προκύπτουν δυσκολίες γιατί δεν μπορούμε εύκολα να ζητάμε επιπλέον πληροφορίες για τα νανοηλικά. Άρα χρειαζόμαστε περαιτέρω προσπάθειες από πλευράς κομισιών για να ξεκαθαρίσουμε πώς καλύπτονται τα ανανοηλικά από το ΡΙΤΣ, Γιατί με αυτό το κείμενο έτσι όπως είναι τώρα, δεν απαιτείται. Δεν απαιτεί από τις επιχειρήσεις α, διανόμου να δώσουν όλες αυτές τις πληροφορίες. Τώρα, για τα υπόλοιπα δεδομένα που δεν είναι ύψιλης ποιότητας και που πρέπει να βελτιωθεί η ποιότητά τους και πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι σπάμε αυτό το φαύλο κύκλο, Κάνουμε αυτή τη στιγμή μία μελέτη που αξιολογεί πώς ερμηνεύει η βιομηχανία ένα συγκεκριμένο άρθρο του Ρίτς ότι θα πρέπει να επικαιροποιεί η βιομηχανία ανατακτά διαστήματα τα ντοσιέ τη. Και μάλιστα κάνουν λάθος ερμηνεία. Ε, συνήθως λένε, καταχωρήσαμε τα στοιχεία, δεν έχουμε επιπλέον πληροφορίες. Όμως αυτό το άρθρο είχε νέα διατάξεις, το αγνοούν. Ε, και οι υπόλοιπε διατάξει του άρθρου λένε ότι τα ντοσιέ αυτά θα πρέπει να επικαιροποιούνται. Θα υπάρξει συμπέρασμα. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται μια εκτελεστική πράξη, ίσως μια αλλαγή στο REACH, για να εξασφαλίσουμε ότι οι επιχειρήσεις παίρνουν στα σοβαρά αυτήν την ιστορία και επικαιροποιούν τις πληροφορίες ανατακτά διαστήματα με νέα επιστημονικά στοιχεία, με νέα δεδομένα, με οποιασδήποτε πληροφορίες απαιτεί η νομοθεσία REACH. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι λάθος το να, μην ξα... αναπληρώνουν άπαξ οι επιχειρήσεις. Είναι λάθος αυτό. Μια και πρέπει να επικυροποιούνται οι... τα ντοσιά αυτά με... επιστημονικά στοιχεία και υπάρχει μια αέναη προσπάθεια, θα πρέπει κάθε 5 ή 10 χρόνια η εταιρεία τουλάχιστον να επικαιροποιεί, α πούμε, μία φορά κατά πέντε, κάθε 5 ή 10 χρόνια και να πληρώνει ένα επιπλέον τέλος. Φυσικά θα πρέπει να το εξετάσει αυτό η Επιτροπή σας, ούτω ώστε να μας βοηθήσει. Να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Να έχουμε ποιοτικά δεδομένα από κάθε άποψη. Διευκρίνησα ήδη το θέμα των περικοπών στο προσωπικό, απάντησα σε αυτό, ε, μας ζητήσαν επίσης να, δουλεύουμε, να δουλέψουμε και αναδρομικά για το θέμα των ενδοκρινικών διαταραχτών. Ε, η Κομισιόν τη ζητήσαμε να μας ε, εκδώσει τρεις ε, ανακοινώσεις που θα οδηγήσουν σε αύξηση προσωπικού για τα φυτοφάρμακα, για την έκθεση, τα όρια, τα όρια έκθεσης στον χώρο εργασίας και τους ενδοκρινικούς διαταράχτες. Έχουμε κάνει δοκιμές και έχουμε αποδείξει ότι εμείς μπορούμε να τα καταφέρουμε πολύ καλύτερα σε αυτά τα παιδεία. Αν χρειαστεί να, δουλεύουμε το 2000, να δουλέψουμε το 2018 πάνω σε αυτά τα τρία θέματα, θα χρειαστούμε επιπλέον προσωπικό. Και αυτό σημαίνει ανακοίνωση από πλευρά τη Κομισιόν με, την, ε, με το δημοσιονομικό δελτίο που τα συνοδεύει αυτά τα κείμενα ούτως ώστε να διευκρινιστούν όλα αυτά, καθώς και το θέμα των κέντρων δηλητηρίας. Εμείς ζητήσαμε από την Κομισιόν να κάνει και μια μελέτη, μάλλον ζητήθηκε να γίνει μια μελέτη για να δούμε ποιες ποια νομοθετικά κείμενα ε, εμπλέκονται όταν βάζουν νέα χημικά οι επιχειρήσεις στην αγορά. Δηλαδή, βασικά βλέπουν τρία ή τέσσερα κείμενα και δεν βλέπουν την πλειάδα των νομοθετημάτων. Καλό θα ήταν να υπάρξει μια μελέτη σκοπιμότητα για αυτό το θέμα, ούτω ώστε οι επιχειρήσει να βλέπουν το δάσο και όχι το δέντρο. Για τη Φιλανδία σε τη διαστολή με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Ποια ήταν τα βασικά ωφέλη. Το θέμα δεν είναι οικονομικό. Είναι το να εξασφαλίσουμε ότι έχουμε τη σωστή υποδομή. Η Φιλανδία, Φερρυπίν, ετοίμασε το κτίριο πριν συσταθεί η ΕΚΑ. Ε, βοήθησε να επιλέξουμε το σωστό κτίριο, προέβλεψε να υπάρχει άδεια για το κτίριο, ούτω ώστε να είναι συνεδριακό κέντρο και να έχει όλες τις εγκαταστάσει που χρειάζεται και παράλληλα ό,τι χρειάστηκε να παραδώσει το φιλανδικό κράτος που εξαρτόταν από το χρόνο το παρέδωσε εγκαίρω, εμπρόθεσμα. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. Αξίζει τα λεφτά που βάζουμε. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο έχουμε και αυτούς τους 10.000 ε, επισκέπτες ε, στη Φιλανδία. Δηλαδή, ε, εμείς βάζουμε αυτό, αλλά η Φιλανδία μας δίνει αυτά που σας είπα. Ε, τώρα θα, θα πρέπει να ψάξουμε για νέο κτίριο, μετά από αυτά τα πρώτα 14 χρόνια, Ελπίζω ότι θα μας βοηθήσει η Φιλανδία, ούτω ώστε να, πάρουμε, να βρούμε το σωστό κτίριο με τη σωστή τιμή. Well, uh, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Δευτά για την παρουσίασή σας, για την επαγγελματικότητα που δείξατε και για την δουλειά που έχετε κάνει τα τελευταία δέκα χρόνια. Σας ευχόμαστε λοιπόν καλή τύχη και καλή συνέχεια. Αγαπητοί συνάδελφοι, παίρνουμε στο επόμενο σημείο. Εξέταση γνωμοδότησης για την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Η Ήτρε κάνει μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας. Συντάκτης της γνωμοδότησης είναι ο κύριος Εκ. Θα του δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο. Κύριε Εκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η μετάβαση από τα ορυκτά καύσιμα σε μια καθαρή πράσινη ενέργεια που είναι κάτι που προσπαθεί και επιζητά η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τεράστιο δυναμικό και πολλά πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα για την κοινωνία, πλεονεκτήματα για τους καταναλωτές και φυσικά πλεονεκτήματα για την οικονομία. Όμως χρειάζεται προσοχή. Χρειάζεται προσοχή για να δούμε ποιος επωφελείται από αυτά τα πλεονεκτήματα και η Επιτροπή μας πρέπει να προσέξει έτσι ώστε τόσο οι καταναλωτές όσο και οι μικρόμες επιχειρήσεις να επωφεληθούν από τις αγορές ενέργειας, να μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν και να χρησιμοποιήσουν λύσεις που θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα, θα μετριάσουν την κλιματική αλλαγή και θα αντικαταστήσουν τα ορυκτά καύσιμα. Τα ορυκτά καύσιμα τα οποία συνεχίζονται να επιχορηγούνται. Γι' αυτό λοιπόν στόχος μας θα πρέπει να είναι η μετάβαση στην πράσινη ενέργεια να γίνει πιο εύκολη στην Ευρώπη. Δυστυχώς στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν πολλοί που δεν έχουν πρόσβαση σε φτηνή και καθαρή ενέργεια. Για το λόγο αυτό χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό κλίμα για καινοτόμες επενδύσεις και τεχνολογία στην, ε, στον τομέα της καθαρής ενέργειας και γι' αυτό χρειαζόμαστε ένα σαφές πλαίσιο νομοθετικό το οποίο θα διασφαλίσει όλα αυτά. Η ενεργειακή μετάβαση επίσης δεν πρέπει να αφορά μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις, δεν πρέπει να είναι μόνο προς όφελος των μεγάλων, αλλά και προς όφελος κυρίως των μικρών. Πρέπει να συνυπολογίσουμε το κόστος της ρήπανσης Τη ατμόσφαιρας υποβάθμιση του περιβάλλοντος και των δαπανών υγεία που προκύπτουν από την εξόριξη και την καύση ορυκτών καυσίμων. Το βάρος αυτό της υποβάθμισης του περιβάλλοντος δεν το επομίζεται η βιομηχανία αλλά η κοινωνία. Γι' αυτό οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα είναι μεγάλο εμπόδιο για την επίσπευση ε, της ενεργειακής μετάβασης για να περάσουμε στην καθαρή ενέργεια. Γι' αυτό καλούμε την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να αναπτύξουν μία σαφή στρατηγική με ξεκάθαρο χρονοδιάγραμμα για την σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα μέχρι το 2020. Ε, θα χαρώ πολύ να ακούσω τους συναδέλφους, τους και ηγητές και όλους εσάς την ανταλλαγή απόψεων που θα ακολουθήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Εκ. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στους ε, σκιώδης Ο κύριος Λαβία έχει το λόγο πρώτος. Ευχαριστώ. Παρεμβαίνω εξ ονόματος της κυρίας Πατριτσέλο που σήμερα δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη συνεδρίαση και θα σας διαβάσω το κείμενό της. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποστήριξε την ανάγκη επιτάχυνσης προς μία ανταγωνιστική οικονομία με χαμηλότερη χρήση άνθρακα μέσα στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος. Στόχοι που θα πρέπει να προωθήσουμε με αποφασιστικότητα. Μέχρι τώρα η πολιτική καινοτομία στον ενεργειακό τομέα είχε τονίσει την ανάπτυξη τεχνολογιών, παραβλέποντας το πιο σημαντικό για τους πολίτες, δηλαδή τις ενεργειακές ανάγκες, ε, τη θέρμανση, κινητικότητα και φωτισμό. Σήμερα αναγνωρίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον καταναλωτή που είναι στο επίκεντρο των αποκεντρωμένων ενεργειακών δικτύων για να βρεθούν ανταγωνιστικές λύσεις με χαμηλή χρήση άνθρακα. Χαίρομαι γι' αυτό. Η Επιτροπή στο κείμενό της ε, υποβάλλει ένα φάσμα μέσων για την καινοτομία με χαμηλή χρήση άνθρακα. Γι' αυτό θα ήθελα να προωθηθεί Επενδύσει επενδύσεις σε όλη την αλυσίδα αυτή και ιδιαίτερα να λάβουμε υπόψη τις μικροεπιχειρήσεις ή τους τοπικούς φορείς που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση επίσης. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την χρήση πετρελαίου και άνθρακα αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τους ε, βιομηχανικούς μετασχηματισμούς και να προτείνουμε εναλλεκτικές λύσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της εξόρυξης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ενεργειακή μετάβαση που έχει μεγάλη σημασία για την ε, πολιτική υποστήριξη των κρατών μελών. Το 2050 θα πρέπει να υπάρχει πλήρης απαλυφή της χρήσης του άνθρακα και ε, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η πρόκληση της αναδιάρθρωσης είναι πολύ μεγάλη, αλλά δεν νομίζω ότι έχουν βρει τα, τα κατάλληλα μέσα από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν ε, τεχνικές λύσεις και μιλάμε για ιδιαίτερες ε, θερμικές εγκαταστάσεις στα κράτη-μέλη. Όμως αυτός ο θερμικός μετασχηματισμός είναι ανεπαρκή σε παλαιά κτίρια. Γι' αυτό κάτι θα πρέπει να γίνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ο μετασχηματισμός αυτός προαπαιτεί πολλά κονδύλια έτσι ώστε οι πολίτες να μπορέσουν να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία μετασχηματισμού. Θα πρέπει να προβληθεί συλλογική χρηματοδότηση, λαμβάνοντας υπόψη τους τεχνολογικούς τομείς, αποθήκευση, ηλεκτροκινητικότητα και κατασκευαστικός τομέας. Θα υποβάλω τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και χάρη στη συζήτηση θα προσπαθήσουμε με τους συναδέλφους να φτάσουμε σε μία φιλόδοξη πρόταση που να τη όλοι μέσα στα πλαίσια των ε, δεδομένων και επιθυμιών ε, της Επιτροπής Βιομηχανίας. Ευχαριστούμε τον κύριο τους κυρίους ε, Λαβία και Πατριτσέλο, κύριο Στανασέσκου. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Όπως γνωρίζουμε, το ΙΔΕΣ Μέτρων για την Καθαρή Ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2016 και συμπεριλαμβάνει την πρόταση της Επιτροπής για την Ενεργειακή Απόδοση, η οποία θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο έτσι ώστε να εκπληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση του στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βασίζεται σε ποιοτική ανάλυση και τα αποτελέσματα διαφόρων αναλύσεων και μελετών για την χρήση καθαρής ενέργειας. Και οι δέσμοι μέτρων αυτοί είναι η πρώτη ευκαιρία που έχουν οι Ευρωπαίοι να εναρμονίσουν τους ε, περιβαλλοντικούς τους στόχους με εκείνους της Συμφωνίας του Παρισιού. Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για την επιτάχυνση της ε, δεσμής μέτρων που αποτελεί μέρος όλου του ε, πακέτου, του Winter Package, είναι πάρα πολύ σημαντική. Και πράγματι τα μεγάλα αποτελέσματα απαιτούν και μεγάλη φιλοδοξία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ώστε να δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και καθαρό περιβάλλον όπου θα ζουν οι πολίτες μας. Ο καταναλωτής πρέπει να είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας για τις εκπομπές χαμηλού διοξιδίου του άνθρακα, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενός ε, ανοιχτού συστήματος. Ο καταναλωτής πρέπει να απαιτήσει λύσεις ε, χαμηλού άνθρακα, πρέπει να απαιτήσει ανταγωνιστικότητα και αποκεντρωμένα ενεργειακά δίκτυα, να είναι ο ίδιος επενδυτής και ε, να ηγηθεί της ανάπτυξης. Για να οδηγηθούμε σε μια οικονομία χαμηλού άνθρακα χρειάζεται να κατανοήσουμε πόσο μεγάλη πρόκληση και πόσο μεγάλη ευκαιρία είναι ταυτόχρονα. Η καινοτομία λοιπόν είναι απόλυτα σημαντική. Θα ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν τον εισηγητή που αναδιατύπωσε τις τροπολογι... κάποιες τροπολογίες του έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται οι επιθυμίες για τροποποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων ε, μελών είναι αναγκαίο να προωθήσουμε την καινοτομία, γιατί είναι κάτι ωφέλιμο για τις ε, επιχειρήσεις, κυρίως τις μικρομεσαίες, έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε καθαρές καινοτόμες λύσεις για ε, ασφαλή ενέργεια. Θα υποβάλω λοιπόν τις σχετικές τροπολογίες και ελπίζω οι συνάδελφοι να τις ευρουν τις αρεσκές τους. Ευχαριστώ πολύ και Τανέσκου. Από την ECR ε, υπάρχει κάποιος? Όχι. Φιλελεύθερη? Πράσινη? Ούτε. Η FTD. Θα θέλετε να πείτε κάτι. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Εκ για την παρουσίασή του. Πιστεύω όπως και εσείς ότι θα πρέπει να υποστηρίξουμε την καινοτομία στον τομέα των ανανεώσιμων. Όμως, αν και η έκθεσή σας είναι συνενετική, θα ήθελα να εκφράσω ορισμένες επιφυλάξεις. Καταρχήν, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η βιομηχανία σε αντίθεση με αυτό που αναφέρεται καλύπτει το ενεργειακό κόστος. Μιλάμε για την αρχή ορυπαίνων πληρώνει. Πλαίσιο το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί. Δεν πρέπει να υποτιμήσουμε τις προσπάθειες των επιχειρήσεων. Επίσης, εάν χρειάζεται, ε, ένας επαναπροσανατολισμός σε καθαρότερες ενέργειες θα πρέπει να μην γίνεται συστηματική χρήση δημοσίων πόρων. Χρειάζεται τεχνολογική ουδετερότητα, την οποία θα πρέπει να τηρήσουμε. Και τέλος υπάρχει και ο κίνδυνος διαφυγής άνθρακα, διαρροής, κάτι το οποίο προβλέπεται ε, δυστυχώς, γιατί καταλαβαίνετε ότι τέτοιες διαρροές ε, συνδράμουν στην ε, αποδυνάμωση της Ευρώπης. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θα ήθελαν να παρέμβουν. Ο κύριος Μπάρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να συνδέσω αυτό που συζητάμε τώρα με την αυριανή ψηφοφορία για το ΛΥΛΟΥΣΙΕΦ. Ένα από αυτά που μπορούμε να κάνουμε σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση είναι να χτίσουμε ενεργειακά αποδοτικά κτίρια το, τα ξύλινα σπίτια είναι ενεργειακά αποδοτικά. Σίγουρα βέβαια μπορείς να κατασκευάσεις ενεργειακά αποδοτικά σπίτια και με άλλα υλικά. Γιατί όμως να μην εξερευνήσουμε και άλλα υλικά, θα μου πείτε. Γιατί αυτά άλλα υλικά πολλές φορές έχουν υψηλό κόστος παραγωγής. Έτσι λοιπόν το κόστος αντικατάστασης του ξύλου, ιδιαίτερα όταν αντικαθίσταται με τσιμέντο και ατζάλι είναι κάτι που πρέπει να εξετάσουμε γιατί έχει πιθανώς ε, πολλά ωφέλη. Αυτό, θα... Αυτό που θα πρέπει να μας ε, απασχολήσει είναι να δώσουμε ε, προσοχή στην τόνωση της βιομηχανίας ξυλίας διότι οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα είναι χαμηλότερες από ε, εκείνες της παραγωγής τσιμέντου. Είναι πολύ δύσκολο να ξεπεράσει την ε, ενεργειακή απόδοση του ξύλου, διότι απαιτείται συγκεκριμένη χημική διαδικασία για να, για να παραχθεί το τσιμέντο. Το να αντικαταστήσουμε λοιπόν ε, το χάλιβα και το τσιμέντο με το ξύλο είναι πιστεύω κάτι που θα συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση της κλιματικής αλλαγής και αυτή είναι η σύνδεση και στην αυριανή ψηφοφορία για το ΛΟΛΟΣΙΕΦ υπάρχει συμφωνία πολλών ομάδων. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τον εισηγητή όπου είναι δυνατόν στην γνωμοδότηση να αναφέρει τη χρήση της ε, ξυλίας, του ξύλου, διότι είναι ένα υλικό περισσότερο ε, αποδοτικό ενεργειακά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα δώσω το λόγο στον κύριο Τόλκιντς από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευχαριστεί τον ε, κύριο ΕΚ για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, που αφορά την επιτάχυνση της καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας. Οι προτάσεις ε, που υπέβαλε ο κύριος ΕΚ είναι συμπληρωματικές με την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα τη βοηθήσουν η πρόσβαση των πολιτών σε λύσεις χαμηλού άνθρακα είναι στο κέντρο των προσπαθειών μας. Οι πολίτες πρέπει να ε, έχουν τη δυνατότητα πρόσβαση σε καθαρή και ασφαλή ενέργεια. Η σημασία των υπηρεσιών και ο σεβασμός της, στους ε, ιδιωτικούς ε, φορείς και τις οντότητες είναι επίσης κέρια σημασίας κατά τη διαδικασία εφαρμογής. Η ανάγκη να καταργήσουμε σταδιακά τα προγράμματα που στηρίζουν την ε, βρώμικη ενέργεια είναι επίσης σημαντική. Πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια αξιολόγηση, να γίνεται παρακολούθηση των επιχορηγήσεων σε ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν γίνει στα πλαίσια του G7 και του G20 για τις επιχορηγήσεις ορυκτών καυσίμων. Είναι λοιπόν αναμενόμενο τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το, τα σχέδια αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής για να εξαλείψουν σταδιακά τις επιχορηγήσεις ορυκτών καυσίμων. τα προγράμματα αυτά συμφωνούν απόλυτα με τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης. Έτσι λοιπόν η στήριξη της καινοτομία στην καθαρή και ασφαλή ενέργεια είναι κάτι ε, που αφορά όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα θεσμικά όργανα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Εκ, θα θέλατε να ξαναπάρετε το λόγο. Όχι. Σας ευχαριστώ πολύ. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής τροπολογιών είναι η 12 Ιουλίου στις 11 το πρωί. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας στις 28 Σεπτεμβρίου. Το λοιπόν ήταν το σημείο 6. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημέρησης διάταξης. Το οποίο είναι η αντίρρηση για τη γενετικά τροποποιημένη σόγια. Θα έχουμε ένα σχέδιο νομοδότησης για προσψήφιση. Έχουμε πολλούς συνεισηγητές. Και καταρχήν θα δώσω το λόγο στον κύριο Σας. Στάς. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε, μαζί με τους συναδέλφους, τους πρασίνους, σοσιαλιστές, ε, γκουε, γευτιντή και ούτω καθεξής, ε, υποβάλαμε αυτή την αντίρρηση που εντάσσεται μέσα σε ένα τελετουργικό. Θα ήθελα να σας κάνω μία εισαγωγή. Ξέρουμε όλοι τον κανονισμό, ο οποίος ορίζει ότι θα πρέπει να αποσυρθούν οι αρνητικοί αντίκτυποι στην υγεία των ανθρώπων και των ζώων. Στις 26 Ιανουαρίου έγινε μία γνωμοδότηση επί του θέματος σε σχέση με τις εισαγωγές. Αύριο θα ψηφίσουμε επί της πρότασης ψηφίσματος και τα κράτη-μέλη ήταν πολύ επικριτικά κατά τη διάρκεια της ε, διαβούλευσης και μιλήσαμε και για τον αρνητικό αντίκτυπο στην υγεία του ανθρώπου και των ζώων. Είπαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες σε σχέση με την αποτίμηση κινδύνου. Γι' αυτό αναφέρουμε στην ε, αιτιολογική σκέψη ε. ε. Μιλάμε λοιπόν και για τα παρασιτοκτόνα και για τα φυτοφάρμακα. Υπήρχαν ε, αρνητικές επιπτώσεις ως προς τους διαταράκτες, και αυτό το είδαμε ιδιαίτερα στους ε, ενδοκρινικούς διαταράκτες και στα έμβρια. Με βάση τον κανονισμό 11, 1107 του 9. Και γι' αυτό το λόγο, ως συνεισηγητές, ε, με αυτή την αντίρρηση θα, να, θα θέλαμε να επισύρουμε την προσοχή στις ε, αρνητικές επιπτώσεις των παρασίτοκτόνων, ιδιαίτερα στις υποανάπτυξη χώρες, όπου εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους ακριβώς επειδή χρησιμοποιούνται αυτά τα παρασιτοκτόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνεται λόγος για τους στόχους της χιλιετίας και τους βιώσιμους στόχους και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ορίσουμε ένα στόχο για την μείωση αυτών των φανάτων και θα πρέπει να δούμε κατά πόσο είμαστε συνεπείς με τους στόχους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ε, αποτίμησή της μίλησε για αυτές τις εισαγωγές αμφίβολων προϊόντων και ουσιών. Με την εισαγωγή αυτού του προϊόντος ε, καθίσταται σαφές ότι η καλλιέργεια θα αυξηθεί και στις τρίτες χώρες με τις αρνητικές επιπτώσεις που περιμένουμε και που αναφέρονται και σε εκθέσεις των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι λοιπόν το ψήφισμα που έχετε ενώπιόν σας και ελπίζω να φτάσουμε σε μία πλειοψηφία και εδώ και στην Ολομέλεια για να αποστείλουμε ένα πολιτικό μήνυμα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική υποστήριξη για την χρήση αυτού του προϊόντος και στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο όπου η Κορεπέρ δεν πέτυχε την πλειοψηφία που θα επιθυμούσε. Ευχαριστώ. Άλλο συνεισηγητή δεν υπάρχει. Ας δώσω το λόγο στους κοιόδους εισηγητέ. Η κυρία Γιούσο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο εισηγητή τη ομάδα μου είναι ο κύριο Φέρνερ. Ζητώ συγγνώμη εξ ονόματό του. Δεν μπορούσε να παραστεί σήμερα θα μιλήσω λοιπόν και θα διαβιβάσω τις ιδέες του για το θέμα αυτό. Υπάρχει δύο θέματα που πρέπει να θέσουμε, ε, όπως και στις άλλες περιπτώσεις. Πρώτον, ε, η Κομισιόν έχει ξεπεράσει τις αρμοδιότητές της. Δεύτερον, υπάρχει επιστημονική αξιολόγηση. Ε, η Κομισιόν ούτε αγνόησε τις επιστημονικές γνώμες, ούτε ξεπέρασε τις, ε, ε τις αρμοδιότητάς της. Ε, υπάρχει, μια, υπάρχει μια επιστημονική γνώμη που δημοσιεύτηκε το Μάρτιο του 2017. Ο εμπειρογνώμονας ε, συμπέρανε ότι ο, η σόγια είναι καλή, ε, όπως και οι άλλες αντίστοιχες σόγες, ε, και, για το, και για την υγεία και για το περιβάλλον. Ε, το 2015 ε, είχαν ε, κατατεθεί τουλάχιστον 15 αντιρρήσεις για το σχέδιο ε, κειμένου, για το σχέδιο κανονισμού. Υπάρχει ο κόντρος που λέει ότι η ΕΦΣΑ θα πρέπει να κάνει επιστημονική αξιολόγηση. Αν η ΕΦΣΑ φτάνει στο συμπέρασμα ότι το προϊόν ε, με γάμα ταφόμικρον είναι ασφαλές με βάση τις επιστημονικές γνώμες, δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως ο εισηγητής θεωρεί ότι δεν είναι σωστός ο τρόπος να εγκρίνονται αυτοί οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί. Εγώ πιστεύω ότι ένα πράγμα είναι τα φυτοφάρμακα και προφανώς πρέπει να αποφεύγονται, ειδικά τα φυτοφάρμακα τα οποία έχουν αρνητική αξιολόγηση για την υγεία και το περιβάλλον και άλλο είναι αυτή η γενετικά τροποποιημένη ε, σόγια και το αν αυτή είναι κακή για την υγεία, για το περιβάλλον. Έχει αποδειχθεί ότι όχι. Και επομένω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα και κάτι άλλο. Ότι εισάγουμε τεράστιες ποσότητες από τέτοιες, τέτοια σόγια γαματαφόμικρον από τρίτες χώρες, γιατί τα, τη χρειάζεται εκτινοτροφία μας. Και τα ζώα τα χρειαζόμαστε. Αλλιώ, αν δεν έχουμε ζώα, θα πρέπει να τα εισάγουμε απ' έξω. Χρειαζόμαστε λοιπόν αυτή την σόγια για να τα ταΐσουμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η διαδικασία αποτίμησης ε, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι από τις πιο αυστηρές. Έτσι έχουμε το κατάλληλο input και είναι εύρωστη έτσι ώστε οποιοδήποτε γενετικός τροποποιημένος οργανισμός ε, την χάνει αυστηρού ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μία ε, σωστή πρόσβαση στην αγορά με βάση την αποτίμηση της ΕΦΣΑ. Και έγινε λόγος για την ε, τοξικότητα, το επίπεδο τοξικότητας και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν επίπεδα υπολοιμάτων σε όλα τα τρόφιμα, είτε αν είναι τροποποιημένα, ε, γενετικός τροποποιημένος οργανισμός, είτε όχι. Ε, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν ε, θανατωθεί, έχουν σκοτωθεί από μία δραστική ουσία που χρησιμοποιείται στο προϊόν. Δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας μίας από τις δραστικές ουσίες. Θα ήθελα να καταστήσω σε ότι οι ζωοτροφές που, την που είναι στο στόχαστρο αυτών των αντιρρήσεων υφίστανται πίεση, δηλαδή τα ζώα με τι πρέπει να τρέφονται. Δεν έχουμε αυτάρκεια στις ζωοτροφές στο Ευρωπαϊκό Στην Ευρωπαϊκή Ένωση εισαγάγουμε ένα 72% των ζωοτροφών και πολλοί από αυτούς που προβάλλουν την αντίρρηση γνωρίζουν ότι δεν μπορούμε να φτάσουμε στην αυτάρκεια. Μιλάνε λοιπόν για την χρήση παρασιτοκτόνων, για τα... μιλούν κατά των ε, βιοκαυσίμων, τη στιγμή που τα χρειαζόμαστε για να μπορέσει να είναι βιώσιμος ο τομέας των ζωοτροφών και επίσης θα πρέπει να να μην αποκλείσουμε και απαγορεύσουμε αποκλειστικά τη γλυφοσάτη που θα μπορούσε να έχει και ολέθριες συνέπειες. Εάν τα κράτη-μέλη δεν έχουν γνωμοδοτήσει θετικά, γιατί δεν υπάρχει το πολιτικό υπόβαθρο, το ίδιο ακριβώς έκανα όταν ε, μιλούσαμε για τα νεονικοτινοειδή τα οποία απαγορεύτηκαν. Δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό μπορεί να προβληθεί ως βασικό επιχείρημα. Μιλάμε για μια ε, ιδεολογία που δεν επιτρέπει τις συμβατικές καλλιέργειες και τα τεχνολογικά στοιχεία και γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχουν οι σωστές νομικές διαδικασίες για να προωθήσουμε αυτό το ζήτημα. Προσωπικά θα ήθελα να πω ότι μετά την δική μου αντίρρηση για τα νέο νοικοτινοειδή μου επιτέθηκαν ε, μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ο τύπος. Δεν είχα κανένα συμφέρον από τον τομέα και ελπίζω να μην ανασυρθεί πάλι κάτι τέτοιο. Και ο οποιοδήποτε γράψει κάτι τέτοιο θα τα ακούσει από το δικηγόρο μου. Κάτι τέτοιο ε, δεν βοηθά τις πολιτικές συζητήσεις που θα πρέπει να προωθήσουμε επί των θεμάτων αυτών. Ίσως υπάρχουν ε, και εκτιμένα συμφέροντα από άλλες ομάδες του αγροτικού τομέα και πολλές φορές ε, εκπροσωπούν και την κοινωνία των πολιτών. Δεν τη βοηθάμε εάν απομακρύνουμε ε, μία άλλη πρωτεϊνούχα καλλιέργεια, την οποία δεν μπορούμε να καλλιεργήσουμε εδώ στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Κάντενμπαχ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα που πήρατε το λόγο. Συγγνώμη που άρχισα και όλα. Ήμουν στην Επιτροπή Γεωργίας και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι η ασφάλεια των τροφίμων, η υγεία και η γεωργία μπορούν να είναι ε, συμβατά. Γι' αυτό λοιπόν και ε, καταλαβαίνω την ε, κυρία Γκέρλινγκ. Ε, εγώ έχω προσπαθήσει να ασκήσω πίεση και υπάρχει μια ομάδα που ασκεί πίεση. Υπάρχει ένα λόμπι που σε μένα βρίσκει πάντα εφοροέδαφος. Τα παιδιά μου είναι, τρο, είναι ε, το θέμα εδώ τρόφιμα. Τρόφιμα που θα φάμε εμείς, τα παιδιά μας και το θέμα λοιπόν είναι πως ε, η ποιότητα πρέπει να είναι ε, ύψιστη. Η παραγωγή τροφίμων που είναι δηλητηριώδη έχει ε, καταστρεπτικές επιπτώσεις όχι μόνο για τους καταναλωτές τους ίδιους αλλά για το περιβάλλον, για ε, το έδαφος, ε, για τα έντομα. Και αυτές είναι οι ομάδες πίεσης που εμένα προσωπικά με ενδιαφέρουν πολύ. Και είναι σίγουρα μια πολιτική απόφαση ενώ θα έπρεπε να είναι βασισμένη σε επιστημονικά στοιχεία. Το όλο θέμα με τη Μοσνισάντο νομίζω πως ε, καθιστά τα πράγματα πολύ σαφή. Έγιναν έρευνες οι οποίες δεν ήταν καθόλου ανεξάρτητες, δεν χαρακτηρίστηκαν καθόλου από διαφάνεια. Γι' αυτό λοιπόν η έγκριση ε, αυτή δεν ε, έγινε από όλα τα κράτη-μέλη. Υπήρξαν κάποια κράτη-μέλη που διατύπωσαν ε, αιτιολογημένες αμφιβολίες και για αυτούς τους λόγους όλους λοιπόν εγώ θεωρώ πως δεν θα έπρεπε να επιτραπεί το DAS 68416-4 γενετικά τροποποιημένη σόγια ακριβώς γιατί παραμένουν πολλά ανοιχτά ερωτήματα ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το φυτό αυτό και τους ε, τρόπους με το οποίο καλλιεργείται. Ε, τα αλλεργιογόνα που περιέχει, τα οποία δίνουν μεν σοδιές πολύ πιο γρήγορα, όμως βάζουν σε κίνδυνο την βιώσιμη ανάπτυξη, το μέλλον και τις επόμενες γενιές. Βάζουν σε κίνδυνο την ποιότητα των τροφίμων που τώρα πολλοί θεωρούμε ως ε, δεδομένη. Γι' αυτό λοιπόν ε, δεν συμφωνώ με την έγκριση αυτή. Δεν συμφωνώ επίσης και με την έγκριση παρόμοιων προϊόντων που στόχο έχουν μόνο το κέρδος και όχι ε, το, καλό, το όφελος του πολίτη και του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Όχι. Κυρία Μπρέτσικη. Από την Κομισιόν, έχει το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Στάς, αγαπητοί ευρωβουλευτές, σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Δεν είναι η πρώτη φορά που σχολιάζουμε το θέμα αυτό από πλευράς μας. Επαναλαμβάνω ότι ακολουθήσαμε όλα τα προβλεπόμενα διαδικαστικά στάδια. Η ΕΦΣΑ έκανε μια πολύ σοβαρή αξιολόγηση κινδύνου και τα κράτη-μέλη σχολίασαν την αξιολόγηση κινδύνου. Η ΕΦΣΑ απάντησε σε αυτά τα σχόλια στη γνωμοδότηση, καθώς και στη μόνιμη επιτροπή, την οποία εγώ, τις οποίες εγώ προεδρεύω. Και κανένα κρατός μέλος δεν αφισβήτησε τη θετική γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Επίσης το κοινό σχολίασε και η ΕΦΣΑ απάντησε στα σχόλια του κοινού, στα σχόλια του κόσμου. Με βάση όλα αυτά και με βάση το γεγονός ότι αυτή η απόφαση ε, σέβεται τον κανονισμό, η Κομισιόν την πρότεινε στα κράτη-μέλη προς ψήφιση. Και όπως πάντα η απόφαση ψηφίστηκε στις 12 Ιουνίου. Δεν υπήρχε καμία γνώμη κατά ε, Η Κομισιόν θα παρουσιάσει την απόφαση στην Επιτροπή Προσφυγών στις 12 Ιουλίου, γιατί δεν υπάρχει ούτε θετική ούτε αρνητική απόφαση. Τώρα, πιο συγκεκριμένα, τα σχόλια. Κατά την άποψη της Κομισιόν, η πώληση της ε, Ένωσης ε, για η συνέπεια για την ανάπτυξη δεν υποσκάπτεται. Καταρχάς είναι μια απόφαση κυρίαρχη μιας τρίτης χώρας να αποφασίσει αν θέλει ή όχι να καλλιεργήσει γάμματα φόμικρον. Αυτό πρέπει να το τονίσουμε. Είναι κυριαρχε αυτές οι τρίτες χώρε. Και δεύτερον, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι όταν εισάγουμε από αυτές τις χώρε, τα πρότυπα τη ευρωπαϊκή Ένωση για την ασφάλεια ισχύουν. Είναι δύσκολο λοιπόν να καταλάβουμε πώς υποσκάπτεται αυτή η πολιτική με τους κανονισμούς που έχουμε για, την, για τους γάμματα φόμικρον. Ε, σε ό,τι αφορά τα προϊόντα προστασίας των φυτών, όπου η σόγια έχει αντοχή. Καταρχάς, υπάρχει χωριστό νομοθέτημα ε, που μιλάει για τα ανώτατα όρια και θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Έπειτα, οι δοκιμές πάντα στον αγρό ε, που γίνονται στους πόρους ε, σόγιας γίνεται για κάθε ένα από αυτά τα φυτοφάρμακα καθώς και για τα φυτοφάρμακα όταν δρούν από κοινού. Επομένως, τα πρότυπα της ΕΦΣΑ πιστεύουμε ότι έχουν γίνει σεβαστά. Και τέλος, η διαδικασία αυτών των φυτοφαρμάκων και τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια δεν ρυθμίζονται στον κανονισμό για τους γάμματα φόμικρον, ρυθμίζονται σε χωριστό νομοθέτημα. Ε, Όμω όταν αυτά τα προϊόντα ε, δηλαδή ε, εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να σέβονται τα μέγιστα όρια καταλήπων. Επίση υπάρχει και ένα άλλο σημείο στο ψήφισμα το οποίο ανέφερα λιγάκι. Ζητήθηκε να αναστείλουμε οποιαδήποτε απόφαση εφαρμογή μέχρι να υποβάλει νέα πρόταση κομισιών. Έχουμε υποβάλει πρόταση, Ούτω ώστε τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να περιορίσουν στην επικράτειά του τη χρήση των ε, ζωοτροφών από γάματα θόμικρων, ορισμένοι μίλησαν για την ε, καινοτομία και για τη βιώσιμη γεωργία. Υπάρχει μια πρόταση επιτάπητος που θα επιτρέψει τα κράτη-μέλη να πάρουν αποφάσεις για τη δική τους επικράτεια, αλλά δυστυχώς αυτή η πρόταση έχει απορριφθεί από το Κοινοβούλιο. Εγώ μπορώ να συνεχίσω τη συζήτηση και θέλω να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Επίση, υπάρχει και μια πρόταση που εκκρεμεί στην Επιτροπολογία, που θα δώσει μεγαλύτερε ευθύνε στα κράτη-μέλη. Συμπερασματικά. Ακούσαμε πάρα πολύ προσεκτικά όλα τα σχόλια και πρέπει να τονίσουμε δεν υπάρχει, ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποσυρθεί το σχέδιο απόφασης. Ε, βασίζεται σε εμπεστατωμένη γνώμη της ΕΦΣΑ. Έχουμε ακολουθήσει και σεβαστεί όλες τις διαδικασίες και τέλος. Θα ήθελα να τονίσω κάτι που υπόθηκε από κάποιον Ευρωβουλευτή, ότι το δικαίωμα ελέγχου του Κοινοβουλίου περιορίζεται στο αν ε, το σχέδιο απόφασης ε, ξεπερνάει τις ε, εφαρμοστικές διατάξεις, τις εφαρμοστικές αρμοδιότητες. Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να δικαιολογηθούμε σε όλα τα επίπεδα. Αλλά ούτως ή άλλως το σημαντικό είναι ε, ότι σας δώσαμε όλες τις εξηγήσεις που θέλατε να ακούσατε και ελπίζουμε με αυτόν τον τρόπο να έχουμε διασκεδάσει τις ανησυχίες σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ όσους συνεισέφεραν και την εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα σχόλια. Θα ψηφίσουμε αύριο για την ένσταση αυτή. Και εάν εγκριθεί στην Ολομέλεια του Σεπτεμβρίου. Περνάμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. μια ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Φέτος η οδηγία για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς έχει φτάσει σε... στα διαναθεώρηση, σε... θεσπίζει μέτρα για την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς και αυτή η ανταλλαγή απόψεων έχει ζητηθεί από την ομάδα ICR και λάβαμε μία επιστολή από τον πρόεδρο της Επιτροπής Γεωργίας, όπου αναφέρεται ότι η Επιτροπή Γεωργίας δεν ε, προτίθεται να ξεκινήσει μία έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας για την αναθεώρηση της οδηγίας. Γι' αυτό σήμερα θα γίνει αυτή η ανταλλαγή απόψεων. Και θα προσπαθήσουμε να ε, είμαστε η επιτροπή που θα ηγηθεί των συζητήσεων. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον κύριο Σετάουσκας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, διευθυντή της ε, Γενικής Διευθυντής ΕΝΤ, που είναι αρμόδια για την πράσινη ανάπτυξη και την κυκλική οικονομία. Κύριε Σαντάουσκας, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.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 της 10 Νοεμβρίου φέτος και να λάβει υπόψη τι εξελίξει των εναλλακτικών λύσεων ε, και τη προστασία των ζώων και επίσης πρέπει να λάβει υπόψη την χρήση των ε, πρωτευόντων ζώων πλην του ανθρώπου στα πειράματα. Αυτό λοιπόν και κάνουμε, γίνεται η αναθεώρηση τη οδηγία και θα σα ενημερώσω σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις. Πριν όμως αυτό θα ήθελα να πω ότι το νομικό πλαίσιο είναι κάπως ατυχές και θα σας εξηγήσω το γιατί. Καταρχάς πρέπει η αναθεώρηση να έχει γίνει το Νοέμβριο. Φέτος όμως τα κράτη-μέλη πρέπει να υποβάλουν εκθέσεις για την ε, κατάσταση εφαρμογή της οδηγία μετά. Έπειτα, ε, μετά την ε, κατάσταση υλοποίηση από τα κράτη-μέλη θα γίνει μία αξιολόγηση το 2019 και η πρώτη στατιστική έκθεση σε επίπεδο ένωσης προβλέπεται επίσης για το 2019. Ε, δεδομένων τούτων λοιπόν μπορείτε να φανταστείτε πως δεν έχουμε πολλά ε, δεδομένα για την ε, υλοποίηση της οδηγίας έτσι ώστε να προβούμε σε αναθεώρηση. Δεν Σταματάω όμω μόνο εδώ. Το θέμα περιπλέκεται περισσότερο με το χρόνο μεταφοράς της οδηγίας στην ε, εθνική νομοθεσία. Το τελευταίο κράτος που εφάρμοσε την οδηγία το έκανε το 2015. Αλλά όπου η οδηγία έχει εφαρμοστεί στην εθνική νομοθεσία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να ελέγξει αν εφαρμόζεται σωστά. Μέχρι τώρα ε, είδαμε ότι 10 κράτη-μέλη έπρεπε να αναπροσαρμόσουν την νομοθεσία του. Τέσσερα από όλα αυτά το έχουν κάνει και τα υπόλοιπα έξι βρίσκονται στη διαδικασία ε, αναθεώρησης και τροποποίηση. Χρειάζεται λοιπόν χρόνο για να γίνουν αυτέ οι αλλαγέ και αυτό δείχνει ότι παραμένουν τα προβλήματα στη μεταφορά της οδηγίας και στις εκτελεστικές διατάξεις. Σίγουρα δεν θα είναι λοιπόν εύκολο να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα της ε, εφαρμογής της οδηγίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαδικασία αναθεώρησης, αρχίσαμε στην αρχή του 2016, συλλέξαμε πληροφορίες ε, από τις αρχές των κρατών μελών, από διάφορες οργανώσεις, από διάφορους ε, δημόσιους φορείς, προστασίας των ζώων μεταξύ άλλων. Εστιάσαμε την ε, προσοχή στην έκθεση αυτή σε τρεις βασικούς στόχους της οδηγίας. Δηλαδή, σε ίσους όρους ανταγωνισμού για όλους τους ε, εμπλεκόμενους φορείς. Δεύτερον, να βελτιωθεί η υγεία και ευζοία των ε, ζώων. Και τρίτον, αύξηση της διαφάνειας οι φορείς που κλήθηκαν να σχολιάσουν τις ε, διάφορες διατάξεις της οδηγίας και να εντοπίσουν αλλαγές που έχουν γίνει στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Και εδώ να πω ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές ε, στα κράτη-μέλη. Εξαρτήθηκε λοιπόν από το στάδιο που είχε φτάσει η οδηγία πριν. Ε, τώρα επιτρέψτε μου να επεκταθώ στους τρεις αυτούς στόχους. Ίση όρια ανταγωνισμού και εναρμόνιση. οι κανονισμοί εναρμονίζουν διαδικασίες, ενώ οι οδηγίες εναρμονίζουν τα αποτέλεσμα. Τα κράτη-μέλη λοιπόν έχουν μια ελευθερία εφαρμογής της οδηγίας στο υφιστάμενο νομικό πλαίσιο. Πρέπει λοιπόν να δούμε τους τομείς όπου υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές αλλά και εδώ θα έχουμε αποτελέσματα μόνο το 2018. Τώρα, βελτίωση της προστασίας ε, των ζώων. Υπήρξαν κάποια καινοτόμα στοιχεία που και η οδηγία, αλλά σε γενικές γραμμές η βελτίωση στην ε, διαβίωση των ζώων είναι ένας από τους κύριους στόχους της οδηγίας, πέραν από την εφαρμογή των τριών R. Έπειτα, πέρα από την αξιολόγηση της ε, καλής διαφύωσης των ζώων, υπάρχουν διάφορες εναλλακτικέ λύσεις για τα πειράματα σε ζώα και εξετάζουμε το στάδιο υλοποίησης των εναλλακτικών λύσεων, εξετάζουμε το στάδιο υλοποίησης και τα αποτελέσματα της οδηγίας και της ε, επικαιροποίηση της διαδικασίας οι εναλλακτικέ λύσεις τώρα που μπορούν να αντικαταστήσουν τη... τα πειράματα σε πρωτεύοντα. Υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι για την υγεία. Χρειάζεται επίσης επικαιροποίηση των στοιχείων για τα πειράματα που γίνονται για, τις, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα και τα νέα φάρμακα. Τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε θα συμπεριληφθούν στην τελική μας έκθεση. Τέλος, ε, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και αύξηση της διαφάνειας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δυνατή μία εις ανάλυση των ε, πρακτικών, των ε, πειραμάτων σε ζώα και των πειραμάτων που δεν γίνονται σε ζώα. Επίσης υπήρξε συνεργασία με πρωτοβουλίες πολιτών που επιθυμούσαν να ε, σταματήσει σταματήσουν τα πειράματα σε ζωντανά ε, ζώα, ή τομές σε ζώντα ζώα. ζώα. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ καλή ε, εικόνα του τι έχει γίνει, τι πρόοδος ε, έχει παρατηρηθεί από την επιστήμη στον τομέα αυτό των πειραμάτων σε ζώα. Τέλος, οι έρευνες των ε, ενδιαφερόμενων φορέων έχουν ολοκληρωθεί. Έχει γίνει μια δημόσια διαβούλευση στο τέλος Μαρτίου, η οποία ήταν ανοιχτή σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Υπήρξαν κάποια προκαταρκτικά ευρήματα και κάποιες προτάσεις έτσι ώστε η τελική έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ε, αντιπροσωπεύει όσο το δυνατόν καλύτερα τα, τις απόψεις όσο το δυνατόν περισσότερων. Παρά λοιπόν το αυστηρό χρονοδιάγραμμα καταφέραμε να έχουμε αρκετά αποτελέσματα. Είδαμε ότι πάνω από χίλιες εγκαταστάσεις χρησιμοποιούν ε, ζώα για πειράματα. Υπάρχουν βέβαια ελλείψεις σε στα στοιχεία, αλλά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα διασφαλίσει όλα τα στοιχεία που θα συλλεχθούν να χρησιμοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και όπως είπα, αυτή τη στιγμή αξιολογούμε τη συνεισφορά των ενδιαφερόμενων φορέων και προσπαθούμε να εντοπίσουμε τα ωφέλη, τις βέλτιστες πρακτικές που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε σε όλη την επικράτεια της Ένωσης και η Κομισιόν θα εγκρίνει την έκθεση μέχρι τις 10 Νοεμβρίου και μετά θα τη συνοδεύσει με ένα έγγραφο εργασίας με συστάσεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, προσβλέπουμε στην ε, συνέχεια της καλής συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θέλουμε και εμείς να συμμεριστούμε τον ενθουσιασμό σας για ε, την βελτίωση των, της διαβίωσης και της προστασίας των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς σκοπούς. Και ελπίζουμε το καλό παράδειγμα να ακολουθήσουν και άλλες χώρες, άλλες περιφέρειες. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη. Η κυρία Γκέρλιν, καταρχήν, γιατί εκείνη έλαβε την πρωτοβουλία για τη συζήτηση αυτή. Ευχαριστώ την Επιτροπή Ήθελα να συζητηθεί αυτό το θέμα, γιατί αυτό το θέμα δεν είναι αποκλειστικής αρμοδιότητας αυτής της Επιτροπής, ούτε καν αυτής της Επιτροπής, αλλά της Επιτροπής Γεωργίας, το θέμα δηλαδή της ευημερίας των ζώων. Αλλά θα έπρεπε να είχε αναλυφθεί μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας γιατί τότε ακριβώς αποδίδουν οι εκθέσεις ίδιας πρωτοβουλίας για να επηρεάσουμε τα πράγματα επί της ουσίας. Δηλαδή να μην προβάλλουμε μόνο ευσεβείς πόθους. Ε, λυπούμε που δεν έγινε κάτι τέτοιο στο Κοινοβούλιο, αλλά ευχαριστώ τους συντονιστές που συμφώνησαν για αυτή τη συζήτηση. Υπάρχουν θέματα τα οποία θα ήθελα να θίξω. Τα περισσότερα έχουν ήδη φυγεί, τα 3R δηλαδή, μείωση, αντικατάσταση και βελτίωση, που έχει προ, θέμα που έχει προωθηθεί και στο Κοινοβούλιο. Και θα πρέπει να σταματήσουμε το ταχύτερο δυνατόν τη χρήση των ζώων στα πειράματα αυτά. Και ε, είχα αναλάβει από την Dagmar Berend αυτό το έργο και είδα ότι υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο έργο και τους ευχαριστώ για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, χαίρομαι που ε, μπόρεσα να μιλήσω και στην περσινή διάσκεψη. Τώρα, ως προς τις βελτιώσεις, υπάρχουν τομείς όπου θα ήθελαν να γίνουν περισσότερα. Ως προς τη χρηματοδότηση καταρχήν. Δυνάμει του άρθρου 48 της οδηγίας αναφέρεται ότι η Επιτροπή και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να προωθήσουν την ανάπτυξη και την ε, επικύρωση ε, πρακτικών και προγραμμάτων. Μόνο 0,4% του συνολικού προεπολογισμού, προϋπολογισμού, δηλαδή 45 δις ευρώ, επενδύθηκε σε εναλλακτικές μορφές και όχι τον πειραματισμό. Και επίσης και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς συμπληρώνεται αυτό το ποσό 0,4%. Δυνάμει του ορίζοντα 2020, 45 δις έχουν αποδοθεί αλλά δεν υπάρχουν εναλλακτικές. Για να μην υπάρχει πλέον πειραματισμό στα ζώα, θα πρέπει να έχουμε πιο στοχοθετημένες επενδύσεις. Τα κράτη-μέλη έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η χρηματοδότηση του ορίζοντα 2020 που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες και επίσης ανταλλαγή απόψεων και πληροφοριών για να φτάσουμε σε πιο ευκτές λύσεις. Θα ήθελα λοιπόν να μας πει η Επιτροπή τι έχει κάνει έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρηματοδότηση για εναλλακτικέ χρήσεις. Υπάρχει και το άρθρο 13 στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ αναφέρεται στις μεθόδους. Δηλαδή, ο πειραματισμός ε, στα ζώα δεν μπορεί να γίνει αν υπάρχει εναλλακτική μέθοδος που αναγνωρίζεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, λυπάμαι, γίνονται συζητήσεις που μου αποσπούν την προσοχή. Οι, τα πειράματα ζώων δεν μπορούν να γίνουν τη στιγμή που υπάρχουν εναλλακτικές, ε, εναλλακτικοί τρόποι. Όμως υπάρχουν κενά που επιτρέπουν σε μερικούς να προβαίνουν σε αυτά τα πειράματα τη στιγμή που δεν υπάρχει ρύθμιση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, υπάρχει δηλαδή μια ανοιχτή πόρτα σε πολλούς τομείς και αυτό δημιουργεί αντίφαση ως προς τη θέση μας. Δηλαδή μπορεί να γίνει ένα πείραμα στη Γαλλία ή τη Γερμανία και μπορεί να γίνει ακριβώς το πείραμα εάν το τελικό προϊόν πουληθεί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν νομίζω ότι αυτή είναι η πρόθεση, αλλά με την αναθεώρηση αυτή θα κλείσουμε αυτό το παραθυράκι. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να βελτιώσουμε τη διαφάνεια γενικότερα. Η Επιτροπή έχει κάνει πολύ καλή εργασία, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε με τη βελτίωση της διαφάνειας, έτσι ώστε να ορίσουμε νέα πρότυπα τάχιστα, έτσι ώστε να λάβουμε υπόψη ότι τα πρότυπα του ΩΣΑ όταν εγκριθούν χρειάζονται πέντε χρόνια μέχρι να, περάσουν στην, ε, να εγκριθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να επιταχύνουμε αυτή τη διαδικασία. Η κυρία Γκροστέτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχουμε μία οδηγία. Η Κομισιόν το φθινόπωρο θα πρέπει να ετοιμάσει μία έκθεση αξιολόγηση τη οδηγία αυτή και διερωτώμεθα μήπω θα πρέπει να την αναθεωρήσουμε ή όχι. Καλό είναι που θέτουμε αυτό το ερώτημα. Πρέπει να υπενθυμίσω ότι αυτή η οδηγία παρά τους τιμητές της δίνει στην Ευρώπη ένα κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που είναι το πιο αυστηρό στον κόσμο σε ό,τι αφορά την προστασία των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους. Και τόσο το καλύτερο που υπάρχει αυτό, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι χρειαζόμαστε, το θέλουμε κάτι τέτοιο. Η οδηγία παράλληλα, μια και είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προβλέπει ε, διοντολογικές αξιολογήσεις υποχρεωτικές πριν περάσουμε σε πειράματα στα ζώα και προβλέπει, όπως είπε η κυρία Γκέρλιν, τον κανόνα των 3 R, δηλαδή την μείωση της χρήσης των ζώων για τα πειράματα, ε, βελτίωση των μεθόδων δοκιμών, ούτω ώστε τα ζώα να υποφέρουν όσο να τρώνε λιγότερο και να αντικαταστήσουμε, δηλαδή να μην χρησιμοποιούμε τα ζώα και να τα χρησιμοποιούμε μόνο όταν δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσεις. Η οδηγία ενθαρρύνει την επιστημονική έρευνα για εναλλακτικέ λύσει, εναλλακτικέ όπω τα πειράματα με ζώα, γιατί είναι σημαντικό γι' αυτό. Και όλοι συμφωνούμε νομίζω εδώ να λάβουμε υπόψη μια ισορροπία ανάμεσα στην ε, ευζοία των ζώων και την επιστημονική πρόοδο. Εν προκειμένου, η Ευρώπη είναι παγκόσμιος πρωτοπόρος ό,τι αφορά τη ε, βιοιατρική έρευνα. Κανένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα ήθελε να χρησιμοποιούνται τα ζώα σαν πειραματόζωα. Είμαστε όλοι, όλοι έχουμε συνείδηση του ότι πρέπει να αποφύγουμε το συντομότερο δυνατόν στην πλήρη απαγόρευση αυτών των δοκιμών. Υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι που αποκαλύπτουμε, που ανακαλύπτουμε σήμερα και θα ήθελα η Κομισιόν να υποστηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις startup ε, που ανα, αναπτύσσουν δοκιμές ε, in silico, που είναι ε, η εναλλακτική λύση. Εγώ τα έχω δει αυτά τα πειράματα. Δεν μπορούμε κάθε φορά να αντικαθιστούμε με αυτές τις μεθόδους ε, τα πειράματα στα ζώα. Όχι κάθε φορά. Αλλά θα καταργηθούν πολλές, ε, πολλά πειράματα με ζώα. Θα μειώσουμε δηλαδή ουσιαστικά τη χρήση των ζώων. Λέω στην Επιτροπή, μα κάνετε ό,τι μπορείτε, ούτως ώστε η έρευνα να μας οδηγήσει σε τέτοιου τύπου εναλλακτικέ λύσεις. Μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ γρήγορα. Έτσι όπως ε, έχει η επιστήμη αυτή τη στιγμή, μου φαίνεται επικίνδυνο και μη ρεαλιστικό να προβλέψουμε την πλήρη απαγόρευση αυτών των δοκιμών, αυτών των πειραμάτων. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ορισμένου τομεί, ε, παραδείγματο χάρη ε, για τις νευρο ε, εκφυλιστικές αρρώστιες, ε, χρειαζόμαστε αυτά τα πειράματα. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε ένα χρονοδιάγραμμα, αλλά όχι ένα χρονοδιάγραμμα για την πλήρη απαγόρευση ε, των πειραμάτων με ζώα από τότε και μετά απαγορεύουμε κάτω 100. Είναι, δεν είναι ρεαλιστικό. Εγώ λέω να κρατήσουμε το χρονοδιάγραμμα τη οδηγία. Όπω είπε και η Κομισιόν μα, υπάρχουν διάφορε ε, δυσκολίε για την ε, ενσωμάτωση τη οδηγία αυτή στην εσωτερική νομοθεσία των ε, κρατών. Πάρα πολλά κράτη-μέλη καθυστέρησαν. Αν είμαστε προθύστεροι, θα δημιουργήσουμε και άλλα προβλήματα. Τώρα που αρχίζει να εφαρμόζεται σωστά η οδηγία, ας περιμένουμε λιγάκι. Περιμένουμε και την έκθεση το φθινόπωρο. Θα πρέπει να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση για την εφαρμογή του κειμένου και για το κατά πόσον σεβόμαστε τους στόχους που τίθενται μέχρι το 2019 και μέχρι τότε να ε, υπάρξει καλή εφαρμογή και με αυστηρότητα εφαρμογή των κανόνων των τριών, άρα αντικατάσταση, μείωση και προσαρμογή. Το να σταματήσουμε κάθε δοκιμή, κάθε πείραμα με ζώα είναι μη ρεαλιστικό. Να μειώσουμε όσο μπορούμε. Α υποστηρίξουμε την έρευνα για να βρούμε εναλλακτικέ λύσει. Α κερδίσουμε χρόνο. Αλλά πρώτα απ' όλα να εφαρμοστεί σωστά η οδηγία και μετά κάνουμε ανατακτά διαστήματα αξιολογήσει και αυτή στιγμή μπορούμε να λάβουμε και άλλε αποφάσει. Τι λαμβάνουμε. Αλλά προ το παρόν νομίζω ότι είναι εντελώ παράλογο να θέλουμε πλήρη απαγόρευση. Thank you very much. Uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκροστέτ. Η κυρία Ντορνανό έχει το λόγο τώρα. Ε, Τον Ιανουάριο μία, ένας οργανισμός προστασίας των ζώων μας έστειλε ένα φιλμάκι για πειράματα στα ζώα σε ένα νοσοκομείο της Γαλλίας ε, και γίνονται πειράματα στο, ε, στον εγκέφαλο αυτών των ζώων για να αντιμετωπιστεί το Alzheimer. Και από ό,τι ξέραμε, ε, τα υπήθηκοι αυτοί ε, στην ουσία ε, είχαν υποβληθεί σε μία διαδικασία αναισθητοποίησης, δεν βλέπουν ποτέ το φως της ημέρας, πολλοί είναι ανάπηροι και έχουν και μεταλλικές, ε, μεταλλικά μηχανήματα στον εγκέφαλο. Βρίσκονται μαζί με γάτες, σκύλους κλπ. Το σχετικό άρθρο ορίζει ότι η Επιτροπή πριν από τις 10 Νοεμβρίου του 2017 με την αναθεώρηση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εναλλακτικέ μεθόδους έτσι ώστε να μην χρησιμοποιούνται ζώα και ιδιαίτερα μη ε, ανθρώπινα πρωτεύοντα. Η Επιτροπή διαθέτει πληροφορίες για νοσοκομεία και εργαστήρια στην Ευρώπη που προβαίνουν σε πειράματα στα πρωτεύοντα εκτός του ανθρώπου και μελέτε σε σχέση με την ανάγκη ύπαρξης αυτών των πειραμάτων, ιδιαίτερα στα πρωτεύοντα αυτά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος. Eichhout. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είχα την εντύπωση ότι σήκωσε το χέρι, αλλά μάλλον το ξέχασα. Να ευχαριστήσω την Επιτροπή, λοιπόν, για τα εισαγωγικά της σχόλια και να κάνω μια ερώτηση ευθύ εξ αρχής. Μιλήσαμε για τις δυσκολίες ε, που θα αντιμετωπίσουμε σχετικά με, την, ε, το πρόγραμμα, με το πώς θα γίνουν τα διάφορα στάδια. Όμως, ε, αν διαβάσουμε την οδηγία, είναι η μόνη αναθεώρηση που προβλέπετε και φέτος δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχουμε. Εσείς πώς ξέρετε ότι σίγουρα θα ακολουθήσει κι άλλη αναθεώρηση στο μέλλον. Γιατί νομίζω πως ε, υπενηχθήκατε κάτι τέτοιο, αλλά εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ε, δούμε να ξεπερνάμε και το 2019. Έχω μία παρόμοια ερώτηση με την Τζούντι Γκέρλινγκ για το άρθρο 13, για τα διάφορα παραθυράκια. Και θα ήθελα μία ξεκάθαρη απάντηση, διότι δεν νομίζω πως χρειάζεται καθόλου πληροφορίες από τα κράτη-μέλη για να δούμε και να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει όντως παραθυράκι στο άρθρο 13, όπου τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν ε, διάφορες εναλλεκτικές μεθόδους, ε, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν, να κάνουν πειράματα και εκτός εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό νομίζω είναι κάτι που δεν μπορούμε να παραβλέψουμε. Μετά, για τα πρωτεύοντα. Υπάρχουν κάποιες συστάσεις στην έκθεση ΣΥΛ αλλά θα συμπεριλάβετε στην αναθεώρηση και τα μη ανθρώπινα πρωτεύοντα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι υπάρχουν μεγάλες ανησυχίες που έχουν εκφραστεί. Και κάτι άλλο, πολύ σημαντικό. Έχουν μειωθεί τα πειράματα σε ζώα. Γιατί το σκεπτικό ήταν να, μειωθούν, να μειωθεί ο ρυθμός των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Και αν δούμε τα στατιστικά στοιχεία για το 2014, μάλλον το 2014 δεν υπάρχουν στοιχεία ακόμα, αλλά από ό,τι φαίνεται τα ζώα που, θα, που χρησιμοποιήθηκαν για πειράματα θα είναι περισσότερα από ό,τι το 2011. Και αν αυτό είναι το συμπέρασμά μας, τότε νομίζω πως είναι προφανές πως πρέπει να γίνει κάτι. Γιατί ο στόχος είναι μείωση, έτσι δεν είναι. Και πρέπει να γίνει αυτό να φροντίσουμε να συμβεί. Έχετε εσείς κάποια, κάποια στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι υπάρχει μείωση και πώς θα διασφαλίσετε αυτό, το να υπάρξει αυτή η μείωση των ζώων που χρησιμοποιούνται για πειράματα. Τέλος, ε, η υλοποίηση των εναλλακτικών λύσεων. Έχω την αίσθηση ότι πολλές φορές η Ευρώπη είναι αργή, διότι πάντα περιμένει την έγκριση του ΑΣΑΜ ένα εναλλακτικό μέτρο που έχει εγκριθεί εντό Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει την έγκριση του ΟΑΣΑ. Πολλέ φορέ περνάνε χρόνια μέχρι να εφαρμοστεί. Πολλέ φορέ περνάνε και 7 χρόνια. 7 χρόνια από τη στιγμή που εγκρίθηκε κάτι εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το περιθώριο πρέπει να στενέψει. Πρέπει να διασφαλίσουμε και εσεί μάλλον ότι από τη στιγμή που συμφωνηθεί κάτι η εφαρμογή πρέπει να γίνεται πολύ πιο γρήγορα από ό,τι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Άλλος? Όχι. Ο κύριος Σαντάουσκας έχει το λόγο. Ξανά. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις ερωτήσεις. Ας αρχίσω λοιπόν με τη χρηματοδότηση. Πράγματι, χρηματοδοτούμε τις εναλλακτικέ ε, μεθόδους εδώ και πολλά χρόνια. Από το πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα 6. Από εκεί ήρθαν τα κονδύλια. Και λόγω του χαρακτήρα της έρευνας αυτής ε, σημαίνει πως ε, χρειάζεται να περιμένουμε πολύ. Οι έρευνες για δερματολογικά θέματα μόνο τώρα έχουν δώσει αποτελέσματα. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν στηρίζαμε ενεργά την έρευνα και την τελευταία δεκαετία η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει παραμείνει σταθερή σε ό,τι αφορά τις εναλλακτικέ μεθόδους. Πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια. Από 35 δισεκατομμύρια το χρόνο, με συγχωρείτε. Βέβαια η βιομηχανία καλλιντικών έχει επενδύσει το δεκαπλάσιο τα τελευταία χρόνια, αλλά στο πρόγραμμα πλαίσιο 7 θα επενδυθούν παρόμοια ποσά. Θα κοιτάξουμε την τοξικότητα διαφόρων χημικών προϊόντων, φαρμάκων, εμβολίων και παρομοίως και για τον ορίζοντα 2020. Θα χρηματοδοτήσουμε 15 ε, διάφορα έργα για τις ε, διαδικασίες ε, in silico και in vitro. Και πρέπει να φροντίσουμε αυτά τα κονδύλια να είναι διαθέσιμα και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεν πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα, όμως εδώ προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες τις ευκαιρίες που έχουμε για να προχωρήσει η έρευνα. Επίσης, χρηματοδοτούμε το Ευρωπαϊκό Εργαστήριο Αναφοράς για τα πειράματα σε ζώα, το οποίο είναι, αν θέλετε, ο κόμβος που ενώνει όλα τα εργαστήρια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το στηρίζουμε με 8 εκατομμύρια ευρώ τους τελευταίους 10 μήνες. Το 2017 ο προϋπολογισμός ήταν 6,5 εκατομμύρια. Μετά θα δούμε, πρέπει να αποφασιστούν ακόμα αυτά ποσά, αλλά νομίζουμε πως η χρηματοδότηση μέχρι τώρα ήταν επαρκής. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν ακόμα τι θα γίνει, όμως από ό,τι βλέπουμε από τα διάφορα εργαστήρια, τις διάφορες εγκαταστάσεις, 38 τον αριθμό σε όλη την επικράτεια της Ένωσης που ελέγχονται από την ΕΚΒΑΜ, μπορώ να πω ότι γίνονται επενδύσεις. Μιλάμε λοιπόν για μεγάλα ποσά. Τώρα, σε ό,τι αφορά το άρθρο 13. Δεν νομίζω πως υπάρχει εδώ κάποιο νομικό παραθυράκι και αν έχουν εντοπιστεί ε, παράνομες πρακτικές, νομίζω πως πρέπει σίγουρα να αντιμετωπιστούν, αλλά δεν μπορείς να κάνεις πειράματα σε ζώα για εξαγωγές. Εάν η νομοθεσία προβλέπει και αναγνωρίζει ε, πειράματα που δεν γίνονται σε ζώα, τότε υπάρχει πρόβλημα επιβολής εάν υπάρχουν στοιχεία για πειράματα σε ζώα εκτός εδάφους ένωσης. Δεν υπάρχει όμως κάποιο νομικό παραθυράκι. Αν υπάρχει και αν προκύψει κάποιο θέμα, το θέμα αυτό θα αφορά μόνο την ε, επιβολή του νόμου. Μετά, η διαδικασία είναι αργή. Αυτό είναι αλήθεια. Και χρειάζεται χρόνος μέχρι να μεταφερθεί στην νομοθεσία των κρατών μελών μέχρι να συμπεριληφθούν όλες οι μέθοδοι του όσα στη μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει διαδικασία επιτροπολογίας, χρειάζεται λοιπόν αρκετός χρόνος. Όμως Ας δούμε τι γίνεται με, τον ε, οργανισμό χημικών που ακούσατε πριν από μία ώρα τον ε, γενικό της να λέει ότι δέχεται τις εναλλακτικέ λύσεις ε, στον κανονισμό ριτς και στα βιοκτώνα. Από τη στιγμή, μάλλον τη στιγμή που εγκριθεί κάτι από τον ΩΣΑ. Δεν είναι υποχρεωτικό να περιμένουμε έγκριση από τον ΩΣΑ, όμως ε, με το να παίρνουμε αυτήν την έγκριση έχουμε μια πολύ καλύτερη εντολή για να προχωρήσουμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μέλη. και του, τα κάθε μέλη και τους φορείς ε, που κάνουν πειράματα σε μια ανθρώπινα πρωτεύοντα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία. Η έκθεση εφαρμογής όμως του 2018 θα τα περιέχει και θα περιέχει τα διάφορα ε, προγράμματα, διάφορα πειράματα που γίνονται σε μια ανθρώπινα πρωτεύοντα. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε μπορούν να μας βοηθήσουν να δούμε ότι υπάρχει μια μείωση στον αριθμό των ε, πρωτευόντων που χρησιμοποιούνται για πειράματα, όμως θα ξέρουμε περισσότερα μόλις έχουμε τα στατιστικά στοιχεία. οδηγία της αναθεώρησης, μάλλον ε, δεύτερη αναθεώρηση της οδηγίας. Δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο, δεν απαιτείται κάτι τέτοιο. Υπάρχουν όμως νομοθετήματα τα οποία θα περάσουν από την άσκηση refit Θα είμαστε λοιπόν επιμελής και ενθελεχείς και σίγουρα θα αξιολογήσουμε όλα τα στατιστικά στοιχεία που θα μας στείλουν τα κράτη-μέλη για το διάστημα 2017-2018. Να σας πω όμως ότι δεν θα έχουμε τα στοιχεία και δεν θα έχουμε τις αποδείξεις πριν από αυτό το διάστημα. Και δεν μπορώ λοιπόν να κάνω κάποια κρίση εκ των προτέρων. Οι προτεραιότητες μα τώρα είναι να διασφαλίσουμε ότι οι πολύ αυστηρέ προϋποθέσεις και να πω εδώ ότι η οδηγία είναι από τις πιο αυστηρές, από τα πιο αυστηρά νομοθετήματα παγκοσμίω που έχουμε εφαρμόσει. Οι πολύ αυστηρές λοιπόν ε, απαιτήσει στις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται τα κράτη-μέλη Εάν εφαρμοστούν, σίγουρα θα μειωθεί ο αριθμός των ε, ζώων που χρησιμοποιούνται σε πειράματα και θα μειωθεί κατά πολύ. Και όπως είπα, εξετάζουμε την μεταφορά της ε, οδηγίας στα κρατη Είμαστε πολύ αυστηροί, εξετάζουμε κάθε λεπτομέρεια, κοιτάζουμε διάφορες έρευνες που διεξάγονται στα κράτη-μέλη. Έχουμε έχουμε περιπτώσεις 25 ε, κράτη-μέλη που έχουν προκύψει προβλήματα, 25 από τα 28. Τα κράτη-μέλη αυτά έχουν ήδη τροποποιήσει κατά πολύ την νομοθεσία τους. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που δεν το έχουν κάνει ακόμα και μία περίπτωση όπου θα ξεκινήσουμε διαδικασία επί παραβάση. Είμαστε λοιπόν ε, ενδελεχείς και νομίζω πως αυτό έχει φέρει αποτελέσματα. Αυτά λοιπόν ε, ως απάντηση στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Um, um, Κύριε Σανταούσκας, για αυτή την ανταλλαγή απόψεων. Ολοκληρώνεται εδώ η ημερήσια διάταξή μας. Θα ξεκινήσουμε αύριο το πρωί στις 9 η ώρα. Καλό απόγευμα, καλούς τριμερείς διαλόγους, ό,τι έχετε.